Possiamo quindi? Anche come componente ci siamo, come numero legale? Possiamo, ok. Buonasera a tutti. Possiamo... Καλησπέρα σε όλους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια συνεδρίαση πολύ πιεσμένη και θα κρατήσει πολύ. Το σχέδιο ημερώσια διάταξη σα έχει αποσταλεί στι 17 Νοεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Την έγκριση των πρακτικών την έχετε στους φακέλους σας. Έχετε και το γλωσσικό καθεστώς στο ενημερωτικό φυλάδιο του Κοκομπού που σας αποστήλαμε. Θα ήθελα να σταθώ για λίγα λεπτά στη σημασία της εξωτερικής ευρωπαϊκής υπηρεσίας της ΕΑΣ ε για τη συνθήκη της Λισαβόνας και στην ανάγκη να παρέμβουμε κατεπηγόντως μέχρι τις, ε, τον Απρίλιο του 2010. Όπω ξέρετε, τα μέλη τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό έκανε και μια ανταλλαγή απόψεων με, τον, με την ε, ύπατη εκπρόσωπο, τη Βαρόνι Άστον. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, όπως έκανα και λίγο πριν ε, στη συνεδρία των συντονιστών, ότι όσον αφορά στη θέση ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα, τι προάλλε ε, έγινε ένα γεύμα, ένα δείπνο εργασία με τον πρόεδρο Μπούζεκ, καθώ επίση και με τον πρόεδρο των εξωτερικών υποθέσεων, τον πρόεδρο Λαμασούρ τη Επιτροπή Προπολογισμών, τον πρόεδρο Αλμπερτίν τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και σε αυτή την περίπτωση υπογράμμισα προφορικός και θα το κάνω και γραπτός ότι η συνθήκη της Λισαβόνα κάνει ακόμα πιο σημαντικό το ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και αυτό για μία σειρά από λόγους. Καταρχάς διότι το Κοινοβούλιο όπως γνωρίζετε πλέον έχει και νομοθετικές αρμοδιότητες και ένα από τα βασικά θέματα με ε, νομοθεσίας που είναι αρμόδιο και το Κοινοβούλιο είναι τα θέματα του προπολογισμού. Και ο προπολογισμό δεν είναι μόνο αρμοδιότητα της Επιτροπής Προπολογισμών αλλά και της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Και από αυτή τη σκοπιά η παρέμβασή μας θα πρέπει να γίνει αμέσως. Το συζήτησα πριν από λίγο και με την Επιτροπή με, ε, με τους συντονιστές ε, για το τι γίνεται με το δημοσιονομικό κανονισμό και την τροποποίησή τους και μία ακόμα πτυχή την οποία θεωρώ εξίσου σημαντική και σε θεσμικό αλλά και σε πολιτικό πλαίσιο είναι το γεγονό ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, είναι δικαίωμά τη και καθήκον τη απονομικής πλευράς να ελέγχει και τα άλλα όργανα, τα άλλα θεσμικά όργανα τα οποία αρχίζουν να ισχύουν με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Μιλάω για την ύπατη εκπρόσωπο, για την ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, την εξωτερική υπηρεσία, γι' αυτό αναφέρομαι και εδώ σε αυτό, ε, και φυσικά συζητήσαμε πριν και για τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Και γιατί είναι σημαντικό να συζητήσει αμέσω η συζήτηση μεταξύ ημών. Γίνονται και οι διαθεσμικέ συμφωνίε. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να έχει εξ αρχή τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή τη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προ τη σημασία και το θεμολιώδη ε, ρόλο της Επιτροπής ελέγχου του Προπολογισμού αρκεί να διαβάσετε το άρθρο 269 της Συνθήκης Λισαβόνας όπου λέει ότι το Κοινοβούλιο νομοθετεί μέσω κανονισμών για τα δημοσιονομικά θέματα που καθορίζουν την, τον προπολογισμό, το ποιο είναι υπόλογο τι και τους ελέγχους. Επομένως αυτό σημαίνει ότι από τώρα και στο εξή θα πρέπει να αρχίσουμε να δραστηριοποιούμεθα και σε αυτό το τομέα και όπω είπα και στου συντονιστέ, έχω πρόθεση από την επόμενη εβδομάδα να αποστείλω γραπτό και στον πρόεδρο και στον πρόεδρο τη διάσκεψη των Προέδρων αυτά τα ουσιαστικά σημεία και τον τόσο σημαντικό ρόλο τη Επιτροπή Κοκομπού. Πριν περάσω τώρα στη συνεδρίαση αυτή καθ' αυτή θα ήθελα να σας πω ότι στο τέλος της συνεδρίας στις μισή θα έχουμε ένα μικρό κοκτέιλ διότι αυτή είναι η τελευταία απογευματινή μας συνεδρίαση πριν από τα Χριστούγεννα επομένως θα μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο και ευχές ε, για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2010. Να περάσουμε τώρα ε, και κάποιες αλλαγές ε, έχουμε στη γραμματεία έχουμε μια νέα βοηθό την κυρία Όφστατ η οποία είναι πλέον μέλος της γραμματέας ε, της Επιτροπής μας της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο της καθώς επίσης και την κυρία Μέρι Μόρναν η οποία έφυγε από τη γραμματεία και την αντικαθιστά κυρία Σύφος Περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, απαλλαγή του 2008, Γενικός Προϋπολογισμός, τμήμα 3 και να δώσω αμέσως το λόγο στο μέλος του ελεκτικού συνεδρίου Κέρστη Λάιτ, αν είναι εδώ. Είναι εδώ. Κύριε Πρόεδρε, εξόδο με μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, αγαπητή Επιτροπή, θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια για το κύριο έλεγχο και τα απορίσματα για την ε, η κοινωνική χρηματοδότηση στο κεφάλαιο 6, θέματα συνοχής. Το 2008 η κοινωνική χρηματοδότηση ήταν 36,6 δις ευρώ, των οποίων 24 ήταν επιστροφές στα κράτη-μέλη, τα υπόλοιπα ήταν προκαταβολές. Υπάρχουν πολύ λίγες επιστροφές στον προπολογισμό του 2008 για το περίοδο του 2007. Συνεπώς, η κύρια πρόοδος στην ετήσια αυτή έκθεση αφορά τις δαπάνες για το, την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006. Το, ε, μελετήσαμε την νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών από τα, τα κονδύλια του 2008, τα συστήματα των κρατών μελών που αναφέρονται σε ανακτήσεις και οικονομικές διορθώσεις και τέλος την ε, τη εποπτεία της Κομισιόν. 57% των προγραμμάτων που ελέγχθηκαν για την περίοδο 2000-2006 Εξ αυτό το 57, συγγνώμη, λέξαμε 170 προγράμματα. 57 προγράμματα δεν είχαν λάθος. Είχαν ε, γίνει σωστά η επιστροφή και δεν είχαν λάθη συμμόρφωσης. Το 2007 αυτή η αναλογία ήταν 46. Αλλά 43% των προγραμμάτων στο δείγμα επηρεάζονται από ένα ή περισσότερα λάθη. Το 42% όλων των λαθών είναι ε, ποσοτικά μετρήσιμα. Με βάση αυτά τα ποσοτικά μετρήσιμα σφάλματα, το συνέδριο υπολόγισε την, ε, ε, τον δίκτυ υπερεπιστροφής πάνω από 11%. Το 11% δεν σημαίνει ότι υπάρχει άμεση οικονομική επίπτωση, είναι ένα τμήμα. Είναι τα ποσά πληρωμών που επηρεάζονται από σοβαρά σφάλματα λόγω των συνθήκων πληρωμής και όπου δεν μπορεί να υπολογίσει ακριβώς το συγκεκριμένο ποσό του συνέδριο. Ένα μεγάλο τμήμα του εκτιμωμένου ε, συντελεστή λάθους οφείλεται σε σφάλματα επιλεξιμότητας, που είναι το πιο κοινό λάθος, στο δείγμα. Σε 41 ελέγχους διαπιστώθηκε αυτό. Οι αιτίε είναι προγράμματα των δικαι... οι δικαιούχοι δεν πληρούσαν τις συγκεκριμένε συνθήκες. Ε, σοβαρή αποτυχία ε, σε κανόνες διαγωνισμών και μπήκαν και κόστη τα οποία, για τα οποία δεν έπρεπε να γίνει η επιστροφή. Οι δύο από τις τρεις πρώτες περιπτώσεις ε, είναι το 80% του σφάλματος. Ένα ιδιαίτερο ε, ενδιαφέρον είναι ο αυξανόμενος κίνδυνος στην δήλωση των μη επιλέξιμων προγραμμάτων. Οι εθνικές αρχές ε, δημιούργησαν νέες δαπάνες ε, σε προγράμματα ή ε, τα υποκατέστησαν με μη επιλέξιμες δαπάνες. Και δεν έγινε εκ των υστέρων έλεγχος από τις Εθνικές Αρχές και το συνέδριο βρήκε ότι αυτά τα προγράμματα προσφέρονται σε ασφάλουν περισσότερο από ό,τι αυτά που έχουν επιλογή με το φυσιολογικό τρόπο. Τελειώνει η περίοδος 2000-2006 και οι εθνικές αρχές πιέζονται να απορροφήσουν τα, κονδύλια της Ένωσης. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να επιστραφούν, να πληρωθούν μάλλον τέτοια κονδύλια σε μη επιλέξιμα προγράμματα. Ε, τα συστηματικά αυτά λάθη και η αναφορά ε, διορθώσεων είναι το πιο σημαντικό φίλτρο για εσφαλμένες επιστροφές. Αυτοί έχουν την ευθύνη να διορθώνουν τα σφάλματα που βρίσκονται από τους ελέγχους ex post και να αναφέρουν αυτές τις διορθώσεις στην Κομισιόν. Το συνέδριο όμως βρήκε ότι αυτά τα συστήματα ε, εν μέρη είναι αποτελεσματικά. Και έχουμε επιτέλους και μερικές πληροφορίες για τη νέα προγραμματική περίοδο. Δηλαδή, για την περίοδο 2007-2013 η Κομισιόν ε, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εποπτεία αποτροπής σφαλμών, σφαλμάτων στις επιστροφές. Δεν μπορούν να γίνουν προσωρινές πληρωμές, δεν υπάρχει έγκριση. Ο έλεγχος έγινε, ε, μάλλον ο έλεγχος μας αποδεικνύει ότι η Κομισιόν ακολούθησε τις διαδικασίες έγκρισης, ωστόσο στην περίοδο 2007-2013 ε, υπάρχουν ήδη προγράμματα τα οποία έχουν δηλωθεί στην Κομισιόν πριν ελεγχθεί το συστήματα ελέγχου. Πάντω είναι ένα κίνδυνο τον οποίο διαπίστωσε το δικαστήριο. τέλο δύο λόγια για τι συστάσει μα. Το ελεγκτικό συνέδριο συνιστά στην ε, ε Κομισιόν να εστιάσει τι ε, κατευθυντήριες γραμμές που δίνει στα κράτη-μέλη σε τομεί όπου υπάρχουν τα περισσότερα λάθη. Ο εντοπισμό και η διόρθωση των λαθών αποτελεσματικά σε επίπεδο κράτους μέλους είναι το σωστό. Να συνεχιστεί ο έλεγχος που στηρίζεται στους κινδύνους των λειτουργικών προγραμμάτων και να υπάρχει αυστηρή εφαρμογή των διορθωτικών μηχανισμών, έτσι ώστε να μην υπάρξουν νέα ασφάλματα από τη διαδικασία αυτή. Βέβαια, αν όλα αυτά δεν οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του συντελεστή σφάλματος, η Κομισιόν ε, και άλλοι αρμόδιοι, μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης του προπολογισμού της Ένωσης, θα λάβουν υπόψη ενδεχόμενο αλλαγή στο σχεδιασμό των δαπανών για την προγράμματα συνοχή στο μέλλον. Έχουμε τώρα, λέει ο Πρόεδρο, τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, Σαμέτσκι, και τον Επίτροπο για την Απασχόληση Κοινωνικά Θέματα Ευκαιρίε, τον κύριο Σπίλα. Σα χαιρετίζω και του δύο. Όποιο από του δυο σα θέλει μπορεί να μιλήσει πρώτο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, πρόσωποι του Ελεκτικού Συνεδρίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο για την παρουσίαση στην ετήσια έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τις ε, ευθύνε τη στη διαχείριση του προπολογισμού και στην εκτέλεση. Πάρα πολύ σοβαρά υπόψη για μένα. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να ελέγχεται και να ε, την χάνει καλή διαχείριση. Το Φεβρουάριο του 2008 Δεσμευτήκαμε στην Επιτροπή σας ε, με το πρόγραμμα δράσης που εγκρίναμε για την ενισχύσουμε την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαθετικές δράσεις. Χάρη στο πρόγραμμα αυτό το πολιετές ε, ελεγκτικό πλαίσιο έχει αρχίσει να δίνει θετικά αποτελέσματα. Η πιο πρόσφατη προσωρινή έκθεση που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2009 περιγράφει τις πρόοδους μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2009 σε ό,τι αφορά τις ε, χρηματοπιστωτικές διορθώσεις 911 εκατομμύρια ευρώ ε, διόρθωσε μέχρι την περασμένη εβδομάδα με αποφάση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια που ε, διορθώθηκαν το 2008, οπότε για τη διετία έχουμε περίπου 2,5 δις ευρώ. Και έχετε τα στοιχεία αυτά στα χέρια σας και μάλιστα και στις οθόνες σημαντική αύξηση σε σχέση με το 1,3 δις που είχαμε διορθώσει στη διετία 2006-2007 πριν τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα δράσης. Με άλλα λόγια, είναι καθοδόν προς διόρθωση 1,2 δις ευρώ. Με την κοινή ε, στρατηγική ελέγχου των ε, διορθωτικών ταμείων θα συνεχίσουν οι γενικές διευθύνσεις στην προσπάθεια να μειωθεί το σφάλμα. Το πρόγραμμα δράσης δεν έχει δώσει ορατό αντίκτυπο ακόμα για το σφάλμα γιατί το 2008 όλες αυτές οι δράσεις έγιναν προηγουμένως πριν τεθεί σε Το 11% είναι υψηλό ποσοστό βεβαίως αλλά φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο προς βελτίωση. Το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι 57% των προγραμμάτων ε, ε, δεν έχουν κανένα σφάλμα ενώ 46% ήταν το 2007 σημαίνει. Ότι έχουν περιοριστεί τα σφάλματα αριθμητικά σε απόλυτους αριθμούς, όπως ήδη είπε η προλαλήσασα, και περιορίζονται σε λιγότερα προγράμματα και σε λιγότερους τομείς. Τι μέτρα λαμβάνουμε για να μειωθεί ε, το ποσοστό του σφάλματος. Θα σας απαντήσω στα εξή σημεία. Πρώτον, γνωρίζουμε που συγκεντρώνονται τα σφάλματα και εκεί εστιάζουμε και τους ελέγχους, τα προγράμματα εκείνα και τα κράτη-μέλη που πλήττονται περισσότερο. Τα σφάλματα αφορούν κυρίως την Κούμβρια και την Καλαβρία στην Ιταλία και στην Ισπανία ορισμένα προγράμματα. Ενώ ορισμένα προγράμματα του Ιντερεγ επίσης ε, αμέσως λαμβάνουμε μέτρα όταν βλέπουμε κάποιες αδυναμίες και όσα σφάλματα εντοπίζουμε παρακολουθούνται και τα κονδύλια ανακτώνται. Γιατί υπάρχουν παρεξηγήσει εδώ και θα ήθελα να τι διασκεδάσω. Ε, οι ε, αριθμίες δεν σημαίνουν πάντα απάτη για τα σταλεία. Το 2008 έγιναν κάποιες δράσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αρκετό. Έχουμε μηδενική ανοχή απέναντι στην απάτη. Στη συνέχεια, έχουμε μια στρατηγική προληπτική για το κλείσιμο των προγραμμάτων 2000 με 2006 και είμαστε πεπισμένοι ότι ε, είναι αποτελεσματική αυτή η στρατηγική. Ε, σύντομα, προσεχώς θα σας φέρει έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, μάλλον θα δείξει ότι το ένα ασφάλμα σφάλμα στο Περιφερειακό Ταμείο για την περίοδο 94 με 2001 είναι στην αρμόδια γενική διεύθυνση. Έχουμε ένα πολιετές πρόγραμμα ελέγχου που περιορίζει σημαντικά το σφάλμα σε σχέση με το ετήσιο σφάλμα που βρίσκει το ελεκτικό συνέδριο. Ε, και για την προγραμματική περίοδο 2000 με 2006 θα μειωθεί το σφάλμα και με χαρά να συνεργαστούμε με το ελεγκτικό συνέδριο. Στη συνέχεια, διασφαλίζουμε ε, μια ομαλή έναρξη τώρα της επόμενης προγραμματικής περίοδου 2007 με 2013 σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Εκ των προτέρων επενδύουμε και έτσι ώστε τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου να είναι αποτελεσματικά ευθύ εξ αρχής. Χρησιμοποιούμε μια μεθοδολογία αντίστοιχη με του ελεκτικού συνεδρίου και τώρα ολοκληρώνουμε ε, τον ε, λογιστικό έλεγχο των δειγμάτων του 2007-2013 για να έχουμε μία ένδειξη για το σφάλμα. Τα πρώτα αποτελέσματα λοιπόν του λογιστικού ελέγχου δείχνουν ότι ο ενισχυμένος έλεγχος για τη νέα περίοδο φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Και ε, είναι κάτω του 5% δείξη του σφάλματος για τα κράτη-μέλη που έχουν βελτιωθεί τα συστήματά τους. Στη συνέχεια, αξιολογούμε τις αιτήσει αξιολογήσεις και τον Οκτώβριο βγάλαμε νέες οδηγίες που καλούν τα κράτη-μέλη να βασιστούν στα συμπεράσματα ε, και να ε, προστρέξουν στη βοήθεια που τους παρέχουμε. Το 2010 θα αναθεωρηθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός και έτσι θα ενισχυθεί η νομική βάση για αιτήσει συνόψεις και περιλήψεις και προσβλέπουμε συνεργασία μαζί σας για να ε, ενισχύσουμε τη λογοδοσία και τη τα λογιστικά των κρατών μελών. Τέλος, το 2009 έχουμε κάνει και δράσεις προς την απλούστευση. Ο Επίτροπος κ. Σπίτλα θα σας ενημερώσει εκτενέστερα για το θέμα αυτό. Συμφωνώ απολύτως με τις συστάσεις του Ενεκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή του και όλοι βεβαίως εφαρμόζουμε αυτά. Έχουμε θέσει σε ισχύ όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ε, έχουμε μηχανισμούς ε, συνοχής ε, αποτελεσματικούς με μείωση του σφάλματος. Μέχρι τώρα οι ενδείξεις μας λέγουν ότι πηγαίνουμε όντως στη σωστή κατεύθυνση και θα ακολουθήσουμε την κατεύθυνση αυτή μέχρι να αποδώσουν πλήρως τα μέτρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. τον Επίτροπο. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Επίτροπο Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας μιλήσουμε σε αυτή την Επιτροπή. Ο συνάδελφός μου, Επίτροπος Σαμίτσκι, σας ε, έκανε μια σύνοψη των βασικών σημείων και των βασικών ε, κατευθυντήριων γραμμών των δραστηριοτήτων μας και της ε, ανταπόκρισης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα εστιάσω στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης της με στόχο να βελτιώσει περαιτέρω την ε, διαχείριση και την εποπτεία των ε, κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό έγινε για να έχουμε και συστάσεις από την ε, δική σας επιτροπή και ως τμήμα του προγράμματος δράσης θέλουμε να διασφανίσουμε ότι η αναστολή των πληρωμών και οι διορθώσεις οι διορθώσεις θα εφαρμόζονται πιο αυστηρά. Στην τελευταία έκθεση το ελεγκτικό συνέδριο αναγνωρίζει πολύ σημαντική αύξηση τόσο των ε, ε, ε, αναστολών όσο και των διορθωτικών διαδικασιών. Ο κύριος Αμέτσκι μόλις σας ενημέρωσε για τη συνέχεια της πολιτικής ευθύς και το 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας έδωσε και τα σχετικά στοιχεία. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σε σχέση με τις προηγούμενες αιτήσεις εκθέσεις, είχαμε κάποιες πολύ σημαντικές θετικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, το Ελεκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι είχαμε μόνο εννέα σφάλματα ε, στα 49 σχέδια τα οποία παρακολουθήσαμε και από αυτά τα 9 μόνο 4 θεωρούνται ε, ότι μπορούν να ποσοτικοποιηθούν από το ελεκτικό συνέδριο και θεωρούν ότι έχουν κάποια οικονομική επίπτωση. Άρα, οι αιτήσει εκθέσεις δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθυντών περιλαμβάνουν μια πάρα πολύ σωστή και πολύ καλά στοχευμένη εκτίμηση των προγραμμάτων υψηλού κινδύνου και των κρατών μελών. Ωστόσο είναι σαφές ότι το συνολικό ποσοστό σφαλμάτων που διαπιστώνει το, συνέδριο, το Συμβούλιο συγγνώμη, εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και ο τελικός στόχος του προγράμματος δράσης είναι να μειώσουμε αυτό το ποσοστό. Ο κύριος Σαμέτσκι μόλις σας ε, εξήγησε τι δράσεις ε, έχουμε αναλάβει για αυτό το σκοπό. Ε, έχουμε και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας ακόμα καλύτερα. Δύο από τις βασικές ε, προληπτικές δράσεις αυτή του νέου πλαισίου περιλαμβάνει την εκ των προτέρων ε, αξιολόγηση για τα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών και δεύτερον να υπάρχουν στρατηγικές ε, ελέγχου για κάθε πρόγραμμα. Το 2008 και το 2009 τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκαναν πολλές προσπάθειες για να ε, εισαγάγουν αυτό το σύστημα σωστά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σκοπεύει να τηρήσει αυτό που της ζητεί το ελεγκτικό συνέδριο, δηλαδή να απλουστεύσει με προσεκτικά. Simplify with care και επίσης ε, θέλει να εφαρμόσει ένα πλουστευμένο δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2007 και το, έως το 2013 και για τις διοικήσεις και για όσους λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η δυνατότητα να ε, δηλώνονται το έμεσο κόστος ε, σε, υπήρχε από την αρχή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Χαίρομαι που σας επισημαίνω ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν αυτή τη διαδικασία απλούστευσης. Ελπίζω ότι η απλούστευση αυτή θα επεκταθεί και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, και τι τροποποιήσει που κάναμε το 2009. Επίση, εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονε από τα κράτη-μέλη για τι διατάξεις αυτές. Ε, όσον αφορά τώρα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού που συζητάτε αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, θεωρούμε ότι Έχουμε κάνει όσο το δυνατόν περισσότερες απλουστεύσεις ε, μέχρι τούδε χωρίς να ε, ασφυζητήσουμε καθόλου τη βάση του ε, πλαισίου διαχείρισης από το 2007 στο 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εφαρμόζεται στα πλαίσια μιας πολύ μεγάλης κοινωνικής κρίσης ε, και η βοήθεια που παρέχει το Κοινωνικό Ταμείο στους ευάλωτους, κυρίως στους ανθρώπους που έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους, είναι μια υπενθύμηση και μάλιστα πάρα πολύ εύστοχη του ε, ρόλου της Ευρώπης ως κοινωνική Ευρώπη της αλληλεγγύης. Ένας λοιπόν από τους ρόλους της διαχείρισης θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική αλληλεγγύη. Γι' αυτό ακριβώς και θεωρώ ότι στους επόμενους μήνες θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά τη μελλοντική οργάνωση αυτής της κοινή διαχείρισης διότι χρειάζεται και ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και του Ευρωπαϊκού Ταμείου, καθώ επίση και να εστιάσουμε περισσότερο στα επιτέχματα που έχουμε υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών, Αυτά λοιπόν κύριε και κύριοι, είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Σπίτλα. Να δώσω το, ρόλο, το λόγο στον uh, κύριο Λιμπεράτσκι για να μας μιλήσει για την απαλλαγή για το 2008. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ένα σύντομο σχόλιο. Έχουμε στα μας δύο πολύ διακεκριμένους επιτρόπους. Βέβαια θα αλλάξουν. Ε. Είναι μια τελευταία ευκαιρία να διδαχθούμε για τα θέματα για τα οποία συζητάμε για το 2008. Πρώτη ερώτηση. Κύριε Επιτροπή, γιατί έχουμε αυτή την ψηλή συχνότητα σφαλμάτων σε σχέση με το 2007, δηλαδή οι μισές από όλες τις πληρωμές, κάθε δεύτερη πληρωμή δηλαδή, δεν είναι σωστή. Όταν το ποσοστό σφάλματος είναι τόσο μεγάλο, πώς μπορούμε εμείς να είμαστε σίγουροι ότι το νούμερο 11% είναι ακριβές όσον αφορά τις ε, οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να είναι παραπάνω από 11%. Η έκθεση επίσης αναφέρεται 33% προγραμμάτων στην παράγραφο 6.17. Αυτή είναι η πρώτη ερώτησή μου κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να κάνω όλες τις ερωτήσεις ή να περιμένω να πάρω απάντηση. Chi vuole rispondere dei commissari? Prego. Ποιος επίτροπος θα απαντήσει, έχετε το λόγο. The frequency of errors, uh, detect... Η συχνότητα σφαλμάτων που εντοπίστηκαν στον έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου μειώνεται σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό είναι γεγονός θετική η τάση. Γιατί είναι ψηλό το σφάλμα σε συχνότητα. Διότι οι πράξεις που έγιναν στο Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά είναι περίπλοκες και αφορούν πάρα πολλούς δικαιούχους και πάρα πολλούς φορείς. μέσα στην αλυσίδα λοιπόν αυτή των πράξεων συμβαίνει. Μερικοί άτομα ή όργανα κάνουν λάθη. Okay, the second question would be... okay, δεύτερη ερώτηση για το 2006. Το σφάλμα 12% αντιστοιχεί σε 4 δις ευρώ. Το 2007 11% είναι Πέντε δις. Ποιο είναι το ποσό για το 11% για το 2008. Είναι 2,7, είναι 4, τι είναι. Και είναι η αλήθεια να προσθέσουμε αυτά τα ποσά προκειμένου να έχουμε ένα σύνολο, τη συνολική εικόνα για τα τρία χρόνια. Δηλαδή να προσθέσουμε όλα μαζί τι μας δίνουν, 12 μας δίνουν, ναι. δις, 14 δις, τι μας δίνει. Απάντηση. Δεν συμφωνώ με αυτή την ερμηνεία. Όπως συντελεστή σφάλμα το 2006, 7 και 8 μεταφράζεται σε συγκεκριμένα ποσά. Για το 2008, το 11% ποσοστό σφάλματος προκύπτει από εφαρμογή της μεθόδου του ελεγκτικού συνεδρίου η Κομισιόν δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες. Δεν την αφισβητούμε. επαναλαμβάνω δεν την αφισβητούμε τη μέθοδο. Το 11% είναι μια εκτίμηση ε, κινδύνου σφάλματος στην πολιτική συνοχή από την Κομισιόν το 2008. Αυτό είναι, σαν, είναι ένα στιγμιότυπο. Τραβάμε μια φωτογραφία. Το ελεκτικό συνέδριο όταν κάνει τον έλεγχό του. Αυτό το νούμερο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να υπολογίσουμε οικονομικές διορθώσεις για το 2008. Οι οικονομικές διορθώσεις δεν είναι 11% στην αξία των πληρωμών για το 2008, όπως είπα και πριν, λόγω διάφορων βημάτων στη διαδικασία τα επόμενα χρόνια μερικά από τα ασφάλματα θα εξηγηθούν. Μερικές δαπάνες θα αντικατασταθούν με άλλες δαπάνες όπου δεν θα υπάρχει ασφάλμα. Γι' αυτό το τελικό που θα για το 2008 πιθανότητα θα είναι πολύ πιο κάτω από το 11%. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Τρίτη ερώτηση. Πόσα χρήματα ανακτήθηκαν στο τέλος του 2008 γιατί με τα προγράμματα δράσης η ανάκτηση για το 2000 μέχρι το 2006 μέχρι το 19 το του 1999. Από ποιες χώρες είναι τα πιο μεγάλα ποσά ή πόσο θα έπρεπε να ανακτηθεί μετά το 2000-2006 αλλά δεν έχει ακόμα ανακτηθεί ως ποσό. Well, ε- Απάντηση. Θα επαναλάβω τα νούμερα από τον πίνακα. Το συνολικό ποσό διορθώσεων που ανακτήθηκαν από το Ταμείο Συνεχής και Διορθωτικά 2006-2007 1,3 δις. Οι διορθώσεις μέχρι στιγμής και τα χρήματα που ανακτήθηκαν για το 2008-2009 είναι 2,3 47 δις. Υπάρχουν και άλλες διορθώσεις καθοδόν 1,2 δις. Το σύνολο 2008-2009 θα είναι περίπου 3,7 δις. Τώρα, τα ποσά, τα ανακτηθέντα κατά χώρα Τα νούμερα μας δείχνουν ότι τρεις είναι, μάλλον τα κράτη μέλη από τα οποία ανακτήθηκαν τα μεγαλύτερα ποσά για την περίοδο 2000-2006, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, η τελευταία ερώτηση. Πήραμε τις γραπτές σας απαντήσεις και έχουμε μια θέση για την έρευνα και ανάκριση 224 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι πολλά τη στιγμή που συζητάμε για δισεκατομμύρια δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, η ενάκτηση, είναι 3,7 δις ή εκατομμύρια. Τέλος πάντων. Ερωτώ, τι πρόοδος έγινε στην κοινή παρακολούθηση των δαπανών για εξωτερικές δράσεις. Διότι είχαμε μια καλή έκπληξη, η συχνότητα λαθών, που ήταν πριν 70%, τώρα είναι γύρω στο 45%. Μεγάλη πρόοδος. Πώς έγινε αυτό. Prego. μου rispondete. The first, uh, the, the first piece of reply... Απάντηση. Πρώτη απάντηση. Ο πίνακας που δώσαμε στις γραπτές απαντήσεις το νούμερο είναι σε εκατομμύρια, αλλά το 3,9 που ανάφερε είναι 3,9 δι ευρώ. Τώρα για τις εξωτερικές δράσεις, δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά, για τις εξωτερικές δράσεις αυτό αφορά, είναι θέμα που αφορά άλλους επιτρόπους. Εγώ δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Οι εξωτερικές δάσεις δεν είναι στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι στο χαρτοφυλάκιο σας, αλλά επ' ευκαιρία, επειδή ήταν το δεύτερο πιο ευαίσθητο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, ας δώσω και στους άλλους συναδέλφους την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, παρόντες επιτρόπους ε, αλλά και να τους επενέσω γιατί βελτιώθηκαν σημαντικά τα νούμερα. Αυτό ισχύει και για τους δύο τομείς και για την αρμοδιότητα κυρίως του κυρίου Σπίτλα. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μας έχει δείξει ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα με μια εξαίρεση που είναι το Βέλγιο και θα επανέλθω σε αυτό. Το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει διαφορετική μεθοδολογία. Στη διαφορά ανάμεσα στο στιγμιότυπο, το snapshot που είπατε και του ελεκτικού συνεδρίου και της δικής σας ε, μακροπρόθεσμης ανάλυσης. Αλλά μπορεί κανεί να κρύβεται πίσω από τι διαφορετικέ μεθοδολογίε γιατί βγαίνουν διάφορα νούμερα και μπορεί ε, κάποιο να χρησιμοποιεί σαν πρόφαση ότι αν ναι, ξέρει άλλη μέθοδο ακολούθησε αυτό γι' αυτό έχει αυτό το αποτέλεσμα, εγώ έχω άλλο. Ειδικά όταν μιλάτε για 0,11% κύριε Σαμέσχη όπου υπάρχει υποψία απάτης, ε, παρά όλα αυτά είναι 57 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό, έτσι. Είναι λεφτά. Καλό θα ήταν λοιπόν κάποια στιγμή να συζητήσουμε για μια κοινή μεθοδολογία. Δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε σαφή κοινή μεθοδολογία για να κάνουμε το εξή. Να ε, ανακαλύπτουμε, να αποκαλύπτουμε τα ονόματα και να ε, υπάρχει και ένας ας πούμε διασυρμός, μια διαπόμπευση. Μόνο αυτό το naming and shaming πιάνει. Αυτό το κάνει όλο και περισσότερο το Ελεκτικό συνέδριο και το κοινοβούλιο, σιγά σιγά τολμάει να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τελικά βελτιώθηκαν οι αριθμοί. Όταν δεν έχεις ε, κατήγορο και δεν έχει και πρόστιμο να ε, κινδυνεύει να πέσει, τότε τα κράτη-μέλη θα συνεχίζουν ε, όσα έκαναν και στο παρελθόν. Αυτό είναι λοιπόν ο σωστό δρόμο. Ε, χρονικά λοιπόν, πότε βλέπετε μια τέτοια πιθανότητα πραγματικά κοινή μεθοδολογία. Επίση, όλοι διαπιστώσαμε, κύριε Σαμέτσκι, γιατί μιλήσατε για τις αιτήσει ε, συνόψεις, ότι δεν επαρκούν. Πριν από ένα μήνα είχαμε μια ακρόαση εδώ, όπου και πάλι αποδείχθηκε ότι έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα οι αιτήσει αυτές ε, περιλήψεις. Πότε να υπολογίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει και άλλη πίεση στα διάφορα κράτη-μέλη έτσι ώστε όλοι να κάνουν την εθνική ε, δήλωση διαχείρισης και να την υπογράφουν. Οι κάτω χώρες είναι καλό παράδειγμα. Παρακαλώ, θα ήθελα την αίσθησή σας πότε περίπου υπολογίζετε να έρθουν και τα υπόλοιπα. Και προς εσάς κύριε Σαμέτσκι, έχω το εξή ερώτημα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε δοκιμαστικά ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε μια μικρή περιφέρεια, έστω και μικρή γερμανική περιφέρεια, με κοινή μεθοδολογία σε συνεργασία με τις ε, εθνικές και ακόμα και περιφερειακές αρχές για να το δοκιμάσουμε πώς λειτουργεί αυτό. Εγώ θα σας προσέφερα, ας πούμε, το κρατήδιο του Σάλαντ που είναι αρκετά ε, εύκολο λόγω μεγέθους. Ε, ε, γιατί, τι γελάτε. Ε, ένα εκατομμύριο κατοίκους έχει. Και πολλοί είναι οι πόροι που έρχονται από τον προπολογισμό του κυρίου Σαμέτσκι μπορούμε πολύ ωραία να το ελέγξουμε. Και συγκεκριμένη ερώτηση προς τον Επίτροπο κύριο Σπίτλα. Προβλήματα εμφανίστηκαν στο δικό σας τομέα αρμοδιοτήτων, εντάξει πάρα πολύ λίγα, στη Σουηδία πολύ λίγα, αλλά κυρίως στο Βέλγιο. Στη Βαλονία και στο ΕΝΟ της Βαλωνίας ένα πρόγραμμα που εσείς χρηματοδοτήσετε υπήρχε πρόβλημα. Ερώτηση συγκεκριμένη. Πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό το περιστατικό. Τι κάνουν οι υπηρεσίες σας για να επεληθεύσουν ότι δεν έχουν ε, δαπανηθεί σωστά τα κονδύλια ή ότι υπάρχουν ατασταλίες και, αν και απάτες. Αν μπορέσετε να μας το εξηγήσετε. Παρακαλώ. Το... Η παρακαλώ. Well, um, Νομίζω ότι το θέμα της κοινή μεθοδολογίας και το επιχείρημα που παρουσιάζεται είναι πολύ λογικό και με χαρά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου τα δύο αυτά συστήματα να είναι όσο το δυνατόν ε, πιο κοινά και πιο ομογενειοποιημένα. Δράτω με δίκη της ευκαιρίας για να σας εκφράσω και την ελπίδα μου να μπορέσει να συμμετάσχει και το ελεκτικό συνέδριο στην διαδικασία που σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε του χρόνου με μια αξιολόγηση ε, των δαπανών που θα σχετίζονται με την περίοδο 2007-2013 για να επαληθεύσουμε αν αυτός ο νέος μηχανισμός ε, που έχουμε θέσει σε ισχύ λειτουργεί. Ελπίζουμε ότι θα λειτουργεί βέβαια, αλλά θα θέλαμε ε, με χαρά να συνεργαστούμε και με το ελεγκτικό συνέδριο σε αυτή την κοινή διαδικασία. Όσον αφορά τώρα στη δυνατότητα να κατανομάσουμε συγκεκριμένους, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Σα έχω αναφέρει και κάποιες χώρες και κάποιες περιοχές σε δημόσιε παρεμβάσεις μου. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να το χρησιμοποιήσουμε και πιο ευρύτερα, αν θεωρείται απαραίτητο. Και θα ήθελα επίσης να διαβεβαιώσω την Επιτροπή ότι η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής έχει κάνει πάρα πολλέ προσπάθειε για να βελτιωθεί η απόδοση των κρατών μελών σε θέματα διαχείρισης και ελέγχων η Γενική Διεύθυνση οργάνωσε και μία σειρά από σεμινάρια κατάρτισης για τις ε, διοικήσεις και για όσους συμμετέχουν ε, στην μεταφορά κονδυλίων. Έχουν δημοσιεύσει και πάρα πολλές κατευθυντήριες γραμμές ε, και σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να δίνουν μια καλύτερη κατανόηση των κανόνων και των διαδικασιών από τα κράτη-μέλη στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Οργάνωσαν και σεμινάρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για όλα όσα τους αφορούν στο θέμα αυτό. Και θέλουν να συνεχιστεί αυτό ώστε να είναι διαθέσιμες σε όλους οι πληροφορίε για τις βέλτιστες πρακτικέ σε όλου όσου ασχολούνται με τα θέματα διαχείριση. Ο Επίτροπος Σπίτλε, μήπως θέλει να πει κάτι. Αναφέρατε το πρόγραμμα ΕΙΝΟ. και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τα ασφάλματα τα οποία μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και που διαπίστωσε το ε, ελεκτικό συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έφτασαν τα 170 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό είναι για το Βέλγιο, 88.000 ευρώ και το σφάλμα εκεί προκλήθηκε από τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για άλλες δραστηριότητες οι οποίες δεν συνδέονταν άμεσα με το ε, πρόγραμμα. Το εντοπίσαμε αυτό το λάθος και από εκεί και πέρα ξεκίνησε διαδικασία με τους Βέλγους εταίρους και στη συνέχεια το λάθος διορθώθηκε και το θέμα έκλεισε. Που σημαίνει ότι αυτές οι 88.000 ευρώ διορθώθηκαν το θέμα θεωρείται λήξαν και δεν θεωρούμε ότι χάθηκε το κονδύλιο. Επρόκειται για ένα σφάλμα του συστήματος. Γι' αυτό ακριβώς και εκπαιδεύσαμε τις βελγικές αρχές ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρπριντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τη χώρα μου, την Ολλανδία, η υποστήριξη προς την Ευρώπη δυστυχώς όλο και μειώνεται και κάτι που δεν βοηθάει για να αυξηθεί η στήριξη και η υποστήριξη Ευρώπης είναι ε, τα νούμερα που βλέπουμε και τα αριθμητικά στοιχεία για το Ταμείο Συνοχής. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο. Γενικά πρόκειται για τα ίδια κράτη-μέλη που κάθε χρόνο πέφτουν σε σφάλματα. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε περισσότερη πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ίδια αυτά κράτη για να σταματήσει επιτέλους αυτή η κατάσταση. Και θα ρωτούσα τον Επίτροπο τι δυνατότητες βλέπει ακόμα για να αυξηθεί η πίεση στα κράτη-μέλη, να τους τριμώξουν περισσότερο, ας πούμε, με πάυση πληρωμών Κάτι τέτοιο. Και το άλλο έχει να κάνει επίσης με την υποστήριξη ω προς τους στόχους και τη σκοπιμότητα των ταμείων. Μιλούμε κυρίω για τη χρηστή διαχείριση, αλλά για να υπάρχει υποστήριξη και προς την Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε κάποιους στόχους εκ των προτέρων και να τους πληρούμε κιόλας. Τι σκέφτεται ο Επίτροπος, πώς ε, βλέπει την επίτευξη των στόχων στην πολιτική συνοχή. ευχαριστώ πολύ. Για την πρώτη ερώτηση, το κατά πόσο είναι το να σκηθεί πίεση στι χώρε μέλη ή αν χρειάζεται να έχουμε επιπλέον εργαλεία για πειθάρχηση. Δεσμευόμαστε από τους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Η συμπεριφορά μας είναι η ίδια, ό,τι μας επιτρέπει το νομικό πλαίσιο δεν μπορούμε να διακόψουμε τις πληρωμές αν δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένους λόγους να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ροή κονδυλίων εκτός αν έχουμε έντονα αποχρόντες λόγους για να το κάνουμε. Αν θέλουμε να τηρούμε την νομιμότητα όλων των πράξεων της Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη, πρέπει να ακολουθούμε το δημοσιονομικό κανονισμό. Τώρα το να ασκήσουμε επιπλέον πίεση πέραν αυτού που κάνουμε κανονικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Σωστή ερώτηση η αποδοτική χρήση ας πούμε. Βέβαια πάει πέραν του θέματος νομιμότητα των ε, πληρωμών. Πριν από δύο μέρες, Φερρυπίν, ήμουνα στην έκτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την αξιολόγηση των διαρθρωτικών ταμείων. Κάτι που το κάνει η Κομισιόν κάθε δύο-τρία χρόνια. Μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ανάγκη να αυξηθεί η αποδοτική χρήση των διαρθρωτικών κονδυλίων. Αλλά για να αυξηθεί αυτό, πρώτα-πρώτα Πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς πετυχαίνει τους στόχους του. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε πολιτικές που να μετράνε την απόδοση και να έχουμε ποσοτικούς δείκτες επιτυχίας. Στις τελευταίες εβδομάδες, μήνες που μένω ακόμα ως Επίτροπος, θα προτείνω ορισμένα πράγματα για το μέλλον που θα οδηγήσουν σε πολιτικές που θα είναι βασισμένες περισσότερο στην απόδοση και που να μετράνε και να αξιολογούν την αποδοτική χρήση των κονδυλίων. Συμφωνώ όμως γενικά ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες ως προς το τι βαθμό γίνεται επίτευξη των στόχων. Ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τους δύο επιτρόπους για τις εξηγήσει τους. Όπως μας είπε και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Κάλλας, τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο. Και ήθελα να πω στο ελληνικό συνέδριο ότι εκτιμούμε θετικότατα την έκθεσή σας που είναι καλή βάση για συζήτηση μερικές σκέψεις. Πρώτον, δεν υπάρχει απάτη, πρέπει να το πούμε αυτό. Θέσαμε ερωτήσεις στους επιτρόπους, πήραμε σαφή απάντηση για τα σφάλματα. Όταν το ελεκτικό συνέδριο γράφει ότι πολλά σφάλματα οφείλονται στην πολυπλοκότητα των κανονισμών και η Κομισιόν απαντάει στην παράγραφο 1.37 στα γαλλικά ότι φταίει ο νομοθέτης. Εγώ απαντώ. Η Κομισιόν εδώ είναι συνυπεύθυνη για την παραγωγή πολυπλοκότητας. Όλοι πρέπει να έχουμε επίγνωση το ότι η παραγωγή πολυπλοκότητας πρέπει να πάψει. Μιλάμε λέμε φταίει το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο γιατί θα μαλώνουμε μεταξύ μας συνέχεια. Να έχουμε επίγνωση το ότι πρέπει να πάψει αυτή η πολυπλοκότητα, γιατί οι πολίτες δεν αντέχουν πια. Στην έρευνα Φερρυπίν, και το συζητήσαμε με τον αρμόδιο επίτροπο, η Ένωση ε, γίνεται όλο και λιγότερο δημοφιλής λόγω ακριβώς αυτού του χαρακτήρα. Τώρα, ο δείκτης 11%. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Είναι λεφτά που χάθηκαν ή είναι ο αριθμός των σφαλμάτων. Θα μπορούσε κάποιος επίτροπος να μας πει χάσαμε τα χρήματα, δηλαδή το 11% της βάσης 2,5-2,7 δις ή είναι ποσοστό σφάλματος. Το ηλεκτρικό συνέδριο καταλέξει. Αυτό που λέει μας δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι λεφτά που χάθηκαν. Και προτείνω κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω τι λέει το Ελληνικό Συνέδριο και η Επίτροπε, μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια ειδική έκθεση για όλη την οικονομική περίοδο 2000-2006 για να ξέρουμε συνολικά πόσα λεφτά χάσαμε με βάση τις οικονομικές διορθώσεις που κάνει η Κομισιόν και οι κυβερνήσεις Δηλαδή, από τη συζήτηση κατάλαβα ότι υπάρχει το πρόβλημα του ετήσιου χαρακτήρα. Δηλαδή, το ελληνικό συνέδριο υποχρεώνεται από τι συνθήκε να τα βλέπει με ετήσιο πρίσμα. Αν πάρουμε όμω όλα τα έτη μαζί, με διορθώσει που γίνονται καθοδόν, η απώλεια όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης δεν είναι και τόσο μεγάλη. Άλλη παρατήρηση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ρωτήσαμε. Τι λάθη είναι, δώστε μας. Η απάντηση είναι, είναι πολύ λίγα τα λάθη. Αλλά για το ελεγκτικό συνέδριο λέω ότι στη σύνδεξη της γνωμοδότησης για τη συνοχή όταν λέμε ότι η συνοχή επηρεάζεται από μεγάλο συντελεστή λάθους, καλό θα, είναι να πούμε εκτός κοινωνικού ταμείου. Το κάνετε για τη Γεωργία, είπατε. Η Γεωργία δεν επηρεάζεται με εξαίρεση την ανάπτυξη της υπαίθρου, και για το κοινωνικό ταμείο, καλό θα ήταν να κάνετε το ίδιο. Τώρα για τα σφάλματα συνοχής, σφάλματα εκτός κοινωνικού ταμείου. Νομίζω υπάρχει συγκέντρωση των σφαλμάτων, είτε ένα άθροισμα πολλών μικρών σφαλμάτων, είτε συγκέντρωση σφαλμάτων μεγάλων. Και διερωτώ μας προς το 11%. Το 11% είναι σφάλματα 8, 9, 12, 13 έχουν πάρα πολλοί λάθη του 0,5, 0,6 και λάθη 100%. Γιατί υπάρχουν και τέτοια λάθη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την επιλεξιμότητα. Αν έχουμε τέτοια περίπτωση, μήπως υπάρχουν ενώτερες αρχές σε μια χώρα που δίνουν πολιτικές εντολές ένα πρόγραμμα που δεν είναι επιλέξιμο τελικά να γίνει επιλέξιμο. Και μας βγαίνει στο τέλος μετά εδώ το λάθος. Γιατί τόσο μεγάλα λάθη, με 100% ποσοστό λάθος. Το θέμα δηλαδή της συγκέντρωσης και του κόστους. Από τη στιγμή που έχουμε πολύ συγκεντρωμένα σφάλματα, πώς μπορούμε να κάνουμε προβολή στο μέλλον Επαναλαμβάνω, τα πράγματα βαίνουν σχετικά καλώς όπως είπα στην αρχή. Απάντηση. για την ε, περιπλοκότητα της διαχείρισης και τους κανόνες υποπτίας. Η περιπλοκότητα των κανόνων διαχείρισης είναι κάτι το οποίο αυξάνεται με το χρόνο και είναι ίσως ε, αποτέλεσμα των προηγούμενων προσπαθμιών οι κανονισμοί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Η πείρα βέβαια μας δείχνει ότι το πολύ μεγάλο ποσοστό ακρίβειας δεν μας ε, κάνει να αποφεύγουμε τα λάθη. Τους τελευταίους λοιπόν μήνες προσπαθούμε να απλουστεύσουμε τους κανόνες και ως απάντηση στην οικονομική ύφεση και την χρηματοοικονομική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε δύο προτάσεις απλούστευσης των κανόνων των διαθροτικών ταμείων. Ο ένας είναι ήδη ε, σε εφαρμογή και ο άλλος συζητάται τώρα με το Κοινοβούλιο. Και, και στους δύο αυτούς κανόνες, ένας από τους στόχους ήταν να γίνει απλούστερη η διαδικασία και οι κανόνες που σχετίζονται με τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Όσον αφορά τώρα στην αξιολόγηση των σφαλμάτων που έγιναν για την περίοδο 2000-2006, νομίζω ότι μια ειδική έκθεση θα ήταν ιδιαίτερως πολύτιμη και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με χαρά θα μπορούσαν να συνεργαστούν ε, στην εκπόνηση μιας τέτοιας έκθεσης. Θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να υπάρχει η έκθεση αυτή όταν θα έχουν κλείσει όλα τα προγράμματα. Και φυσικά είμαστε διατεθειμένοι και να συνεργαστούμε με το ηλεκτρικό συνέδριο για το θέμα αυτό. Ως προς το ποσοστό σφαλμάτων και το, τη σημασία αυτού του 11% νομίζω ότι προσπάθησα να εξηγήσω τη θέση μου από αυτού και θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προοδεύσουμε είναι να ζητήσουμε από τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου πώς ε, δίνεται η μεθοδολογία και πώς ε, καταλήγουμε στο ποσοστό σφάλματος. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Πίγκλα. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε κάποιες ε, περιπτώσεις για να διευκρινίσουμε το ερώτημα κατά πόσο το ποσό στο οποίο καταλήξαμε μέσω της στατιστικής μεθόδου σημαίνει απώλεια χρημάτων. Το ελεκτικό συνέδριο και οι δύο επίτροποι είπαν σαφώς ότι δεν υπάρχει απάτη στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος. Το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσον το ποσό αυτό σημαίνει απώλεια. Σας ανέφερα την ε, περίπτωση του Βελγίου όπου σας είπα ότι 88.000 ευρώ υπήρξαν αντικέμενο διόρθωσης και επανήλθε, επεστράφει το ποσό στον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυτό δεν ε, προσμετράται ως απώλεια κονδυλίων. Μία δεύτερη περίπτωση που θα μπορούσα να αναφέρω είναι μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, από πλευράς Γαλλίας και εκεί είχαμε ένα ποσό της τάξης των 73.000 ευρώ και λόγω σφαλμάτων ή μάλλον λόγω διαφορετικής ε, μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε στο, ε, χρησιμοποιήθηκε στο σύστημα πληροφορικής έγινε λάθος ε, υπολογισμός ε, στο ποσό της συγχρηματοδότησης. Μετά από κάποιους μήνες βέβαια το λάθος αυτό διορθώθηκε αυτομάτως. Επομένως δεν υπήρχε απώλεια και πάλι, αλλά ήταν ένα ε, σφάλμα το οποίο μπορούσε να ποσοτικοποθεί. Οπότε και πάλι είχαμε λάθος, αλλά δεν χάθηκαν χρήματα. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουμε ποτέ καθαρή απώλεια, αλλά αυτό ε, είναι ακόμα νωρί να το πούμε. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να κλείσουν όλε οι υποθέσει. Όσον αφορά τώρα στην ε, πρόταση να ξεχωρίσουμε τελείως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, νομίζω ότι αυτό θα ήταν κάτι θετικό διότι τα διαρθρωτικά ταμεία αφορούν διαφορετικές ε, αρμοδιότητες. Ακούγεται λογικό αυτό που λέτε, αλλά δεν έχω ακόμα σαφώς διαμορφωμένη άποψη για την απλούστευση. Η δημιουργία ενός νέου συστήματος σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τις πρακτικές ε, πτυχές ε, από την πρώτη στιγμή για να μην είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Ωστόσο, σε αυτή την προσπάθεια πλούστευσης που έχει γίνει μέχρι τώρα, η επιλογή των χονδρικών ποσών για, τα τρέχοντα, για τις τρέχουσες δαπάνες θα σήμαινε στην περίπτωσή μας ότι οι τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις που έχουμε εντοπίσει δεν θα είχαν συμβεί καν εάν είχαμε χρησιμοποιήσει το νέο πλουστευμένο σύστημα των χονδικών ποσών. Ένα άλλο, αποτέλεσμα, ένα άλλο ερώτημα ήταν το θέμα της αποτελεσματικότητας. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε την αποτελεσματικότητα και την απόδοση με διαφορετικές μεθόδους, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε λίγο πιο επιστεμένα αυτό το ερώτημα και αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μία πολύ καλά προετοιμασμένη μεθοδολογία διότι ε, αν είναι, αποτελε... είναι να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να ε, την έχουμε προετοιμάσει κατελήλως. Ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να απαντήσω και εγώ σε κάποια από τα θέματα που έθιξε το... έθιξαν τα μέλη του Κοινοβουλίου το ελεγκτικό συνέδριο όταν κλείσουν υποθέσεις σαφώς θα τις ελέγξει. Το έχει ξανακάνει αυτό στο παρελθόν αλλά χωρίς το μοντέλο διασφάλισης. Το μοντέλο διασφάλισης είναι ένα δαπανηρό ε, μοντέλο το οποίο δεν ε, χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις. Επομένως δεν μπορώ να σας διασφαλίσω ότι θα το χρησιμοποιήσουμε την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε αλλά σίγουρα θα παρακολουθήσουμε το κλείσιμο. Το 11% σαφώς δημιουργεί ερωτηματικά. Πώς καταλήξαμε σε αυτό το 11%. Για να σας το πω απλά, Είδαμε όλα τα προγράμματα των 24,8 δις, ε, ε, κάναμε μια δειγματοληψία 180 προγραμμάτων και από εκεί και πέρα έγινε προβολή αυτών των προγραμμάτων σε όλο το τομέα του προπολογισμού. Ε, χωρίς όμως να περνάμε στα στατιστικά στοιχεία, το, η καλύτερη απόδειξη είναι η σταθερότητα για τον τομέα της συνοχής. Για τα τελευταία τρία χρόνια τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν αντίστοιχα και αυτό συσχετίζεται πάρα πολύ καλά με το γεγονός ότι ελέγχουμε συνεχώς ε, τα ίδια συστήματα και ε, όλα αφορούν την περίοδο του 2000-2006. Αν δούμε ξεχωριστά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να σας υποθυμίσω ότι δεν ε, έχει χαθεί τίποτα εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν τα πήγε και πολύ καλύτερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επομένως, όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία, ίσως μπορέσουμε να εξετάσουμε λίγο πιο ενδιαλοχώς το ζήτημα. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήταν στατιστικά λάθος να ε, ποσοτικοποιήσουμε αυτό τον πληθυσμό των 180 και να καθορίσουμε σαφώς ε, ποσά. Γι' αυτό, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχουμε στοιχεία και για τα δύο ταμεία. Επειδή ε, αυτή τη στιγμή το μοντέλο και για τα δύο ταμεία είναι αντίστοιχο. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας... Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίαση και τους δύο επιτρόπους για τον επικοδομητικό διάλογο που έχουμε μεταξύ ημών και του ελεγκτικού συνεδρίου και των επιτρόπων. Θα ήθελα να ρωτήσω τους επιτρόπους, διότι έχουν και συμπληρωματικέ αρμοδιότητες, αν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο να είναι ζωντανό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, προβλήματα με τα διορθωτικά ταμεία, αν υπάρχουν ε, προβλήματα πριν από το 2000, όταν δεν εφαρμόζαμε ούτε το σύστημα του ε, name and shame, δεν κατανομάζαμε κανέναν, ούτε υπήρχαν τόσο επιστομένοι έλεγχοι. Ξέρουμε όμως ότι υπήρχαν κάποιες χώρες, ακόμα και τότε, που είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα προβλημάτων, για να μην χρησιμοποιήσω πιο σκληρή γλώσσα. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται και ή δυνατόν όσο πιο διεξοδικά γίνεται. Ε, Παραδείγματο χάρη στην περίπτωση του κυρίου Σπίτλα διαπιστώνουμε ότι έγινε μια πάρα πολύ σαφή ερώτηση και λέμε υπάρχει μια περίπτωση στο παρελθόν, στην Ισπανία μάλιστα, γιατί εμείς κάναμε την κάθαρσή μας βέβαια και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πάντα και ελπίζω τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι να εφαρμόζουν τα ίδια γιατί ε, θα πρέπει να εξαφανιστούν τα προβλήματα. Δεν θα σας αναφέρω ποιοι είναι ποιοι, αλλά θέλω να ξέρω τι μας έχει μείνει ως κατάλοιπο από το παρελθόν. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο Σαμέσκη, ο οποίος ε, ανέλαβε και καθήκοντα στα... προς το τέλος της θητείας. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνει για να μας απαντήσει εδώ στην Επιτροπή μας. Παρά το γεγονός ότι αυτά είναι διαχείριση της ε, προκατόχου του. Και πάλι για τις περιπτώσεις που έχουμε πριν από το 2008, είδαμε το 2000-2006, υπονθυμίσαμε κάποιες χώρες, αλλά ξεχάσαμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι τα ποσά όπως παρουσιάζονται θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλη σύγχυση. Για άλλη μια φορά, και αυτή θα είναι τελευταία γιατί μετά θα θυμώσω, έχει πέντε χρόνια που σας ζητάω το ίδιο πράγμα. Όταν μας παρουσιάζονται αριθμητικά στοιχεία για τα ταμεία, για τα προβλήματα, για την ανάκτηση των ποσών, ε, και κάθε φορά κάνετε έκκληση προς τη χώρα μου να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να βελτιώσει τα πράγματα, ε, με συγχαίει λίγο το γεγονό ότι υπάρχουν χώρε που είναι σαν τη δική μου, που έχουν ε, ένα δίστα πάνε και φαίνονται να είναι πιο προβληματικοί και κάποιε άλλε μικρέ χώρε ή και μεγάλες χώρες, οι πιο σημαντικέ όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκριτικά φαίνεται να είναι ε, τα δικά του τα προβλήματα ένα προ πέντε. Επειδή όμω εδώ δεν έχουμε το σύνολο των ταμείων, το σύνολο τη διαχείριση σε κάθε χώρα, εγώ που έκατσα και έκανα του λογαριασμού και είμαι και φιλόλογο και δεν τα καταλαβαίνω και πάρα πολύ καλά αυτά. Αυτό που κατάλαβα όχι από τον πίνακα του κυρίου Σαμέσκη που μας παρουσίασε μόνο ένα-δυο πίνακες, αλλά από τον πίνακα του κυρίου Σπίτλα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρέδωσε αυτό τον πίνακα. Στον τελικό πίνακα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Φτάνει μέχρι το 2006 και δεν υπάρχει το Ταμείο Συνοχής το συνολικό άρθρισμα θα είναι πολύ μεγαλύτερη η σύγκριση. Ελπίζω του χρόνου να μπορέσουμε να έχουμε όλου του συγκριτικού πίνακε, γιατί αν συγκρίνουμε καλά τα πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που μα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνουμε ότι η σύγκριση μεταξύ τη Ισπανία που έχει ένα δι και που είναι ένα ποσό πάρα πολύ εμφανέ και διαχειρίζεται 59.000 ε, δεν ξέρω πόσα μέχρι το 2006 αυτό μου δίνει ένα κλάσμα του 1,48%. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, που εδώ το ξεχάσαμε, το ξέχασε ο Επίτροπος, που διαχειρίζεται ε, πολύ μικρότερο ποσό, φαίνεται μεν πιο διακριτικό το ποσό, αλλά ε, διαχειρίζεται 17 δις και το κλάσμα βγαίνει 0,49%. Υπάρχει προβλήματα, πρόβλημα λοιπόν στο ποιο διαχειρίζεται τι. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να το καταλάβουν λίγο οι πολίτες, να μην τους δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα, διότι έχουμε για πρώτη φορά ε, ακολουθήσει το σωστό δρόμο. Μας παρουσιάζει το ελεγκτικό συνέδριο στοιχεία που δεν προκαλούν σκάνδαλο, δεν προκαλούν αντιευρωπαϊκές τάσεις και σκεπτικισμό Φαίνεται να υπάρχει η καλύτερη δυνατή διαχείριση λοιπόν ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να βελτιωθούν και άλλα τα πράγματα, να ετοιμάζετε τους πίνακες καλά. Γιατί αλλιώς δημιουργείται πρόβλημα. Πάντα ασχολείστε με τον Νότο και πάντα ξεχνάτε κάποιους από τον Βορρά που ασχολούνται με ε, πολύ μεγαλύτερα ποσά και βγαίνουν ποσοστά περίεργα. Σας παρακαλώ μην τα ξεχνάτε. Παρακαλώ. Um, Για τις οικονομικές διορθώσεις από το 1994 στο 1999. Έχουμε κλείσει, έχουμε ε, πάρει όλες τις αποφάσεις μάλλον. Με, περιμένουμε μερικά εκκρεμή σημεία αποφάσεις θα ληφθούν στους επόμενους μήνες με μία επιφύλαξη. Μερικές ε, αποφάσεις έχουν αμφισβητηθεί από οι κυβερνήσεις. Είμαστε σε ευρωδικαστήριο. Οπότε θα χρειαστεί χρόνος γι' αυτό. Όσον αφορά την ακρίβεια των δεδομένων του πίνακα που σας υποβάλαμε, δεν ανάφερε το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι σκόπιμα. Δηλαδή, τα κριτήρια για τις τρεις χώρες είναι ότι οι τέσσερις τρεις χώρες είναι πρώτες όσον αφορά το μέγεθος των διορθώσεων. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τέταρτη χώρα στη σειρά. Η απόσταση μεταξύ των τριών χρονών, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα σας είπα, μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης χώρας, το Ηνωμένου Βασίλειο, είναι μεγάλη η απόσταση. Στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχετικό ειδικό βάρος των διορθώσεων. Ανάλογα δηλαδή με, τις, με τα κονδύλια κατά κράτος την επόμενη φορά αυτό. Και ο Επίτροπος Πίγλα. Σχετικά με το κατά πόσον κλείσαμε την περίοδο 94-99. Κλείσαμε το 94% των προγραμμάτων. 1159 προγράμματα και μας μένουν εκκρεμεί 73. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, πολλοί λόγοι. Ορισμένα θέματα έχουν φτάσει στο δικαστήριο. Οπότε χρειάζεται χρόνος. Τώρα ειδικά για την Ισπανία. Ήθελα να σας πω ότι η ισπανική περίπτωση την ερεύνηση ΟΛΑΦ του 2003 και το θέμα έκλεισε το 2004. Πέρασε στον τύπο πιο πριν, το 2002, και ξανεφανίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου φέτος με την ίδια διατύπωση. Πιθανώς οι δημοσιογράφοι χρησιμοποίησαν παλιά στοιχεία η Κομισιόν με έκανε και μια ειδική μονάδα, task force, για να ερευνήσει το θέμα. Και πρέπει να πετύχουμε μια κοινή συμφωνία με τη συγκεκριμένη χώρα, την Ισπανία, διόρθωσε 105 εκατομμύρια ευρώ και μπλοκάραμε 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Και περνάμε τα μέτρα της κυβέρνησης. Οι διορθώσεις έγιναν το 2004 και 2005. Έχουμε ένα νέο σύστημα χρηματοδότησης, έγινε μια νέα κατάρτιση το 2004 το πρόγραμμα, σημαντικό πρόγραμμα όπως σας είπα που είχε πολλά σφάλματα αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση Επίσης προσοχή δόθηκε και στο πρόγραμμα από τους, ε, την Ισπανική Ελεγκτική Αρχή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι υπό έλεγχο, ελέγχεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και υπευθυνότητα. Επίσης τονίζω, όλα αυτά έγιναν σε πλήρη συνεργασία με τις Ισπανικές Αρχές. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, οφείλω να ομολογήσω ότι η διαδικασία απαλλαγή έχει φτάσει στα όρια της αντοχής της. Ε, οι ερωτήσεις μας έφτασαν ε, χθες το βράδυ στις 7 για απαντήσεις μάλλον. Ε, πολύ λίγο τις μελέτησα δεν ξέρω τι να σας πω. Καλό θα ήταν να έχουμε αν μη τι άλλο 24 ώρες νωρίτερα τις απαντήσεις για να μπορέσουμε να τις μελετούμε και να κάνουμε μια συζήτηση όπως πρέπει. Γιατί έχουμε και νέα ερωτήματα που προκύπτουν. Θα ήθελα να απευθυνθώ και στους δύο επιτρόπους για τα εξή τέσσερα. Η μήνυ δήλωση αξιοπιστίας, μήνυ DAS, που περίπου 4% από το ε, Κοινωνικό Ταμείο προέκυψε με τη νέα διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μας ενδιέφερε γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το δείγμα της Επιτροπής από εκείνο του ελεκτικού συνεδρίου. Και θα ήθελα να μάθω πώς αξιολογούν τα αποτελέσματα και οι δύο επίτροποι και το ελεγκτικό συνέδριο και πώς θεωρεί ότι μπορεί να αξιοποιήσει με αυτή τη μήνυ δήλωση αξιοπιστίας και πώς την αξιολογεί το ελεγκτικό συνέδριο γιατί ακριβώς όταν βλέπω το κοινωνικό ταμείο και τα παραδείγματα του συνεδριού του ελεγκτικού γεννιέται σε μένα η υποψία ότι δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν πάρα πολύ και λυπάμαι για την επιλογή των παραδειγμάτων γιατί δεν έχουν την ε, ισχύ του επιχειρήματο που θα θέλαμε και την πυθό. Δεν Και δεύτερη ερώτηση αφορά την Ελλάδα. Βλέπουμε από τον τύπο ότι η Ελλάδα έχει δείξει δημιουργικότητα στην ε, παραποίηση των στατιστικών. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τα περιφερειακά ταμεία και τα κοινωνικά ταμεία. Τι είναι αυτό που πείθει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τώρα τα στατιστικά στοιχεία και το υλικό που συλλέγει η Ελλάδα είναι το σωστό. Γιατί από ό,τι φαίνεται στον Επίτροπο για την Οικονομία και τα Νομισματικά φαίνεται ότι δώσανε λάθος στοιχεία. Εσάς τι να κάνει να πιστεύετε ότι η Ελλάδα δίνει σωστά στατιστικά στοιχεία για τα περιφερειακά κονδύλια. Για την Ισπανία τώρα και για την έκθεση της συνοχής. Μας κάνει εντύπωση ότι η Ισπανία είναι εκείνη ε, η χώρα συνοχής που υπερέχει ε, στην επιτυχία γιατί από ό,τι φαίνεται είναι στο 105% της Ευρώπης των 27, άρα θα πρέπει να βγει από τη συνοχή. Και τι σημαίνει αυτό, από τη στιγμή που θεωρείς χώρα συνοχής και το χρειάζεσαι ή δεν το χρειάζεσαι, το παίρνει για πάντα αυτό το κονδύλι το περιφερειακό, γιατί η συνοχή σημαίνει να βοηθούμε τις χώρες που χρειάζονται τη βοήθεια και όταν στατιστικά πλέον δεν τις χρειάζονται τις ενισχύσεις, Μήπως θα πρέπει να ε, σταματήσει η επιδότηση. Όχι ότι θέλω πίσω τα χρήματα, απλώς άλλη κατανομή. Άλλη ερώτηση. Και σε ό,τι αφορά τη Γερμανία και σε ό,τι αφορά την Ισπανία, τα μεγαλύτερα προβλήματα τα έχουμε στις δηλώσεις ατασταλιών. Δηλαδή με ποιο τρόπο γίνεται η καταγγελία ή η δήλωση. Αυτό διακυβεύεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει κάνει λοιπόν έτσι ώστε η δήλωση, κοινοποίηση των ατασταλιών και των προβλημάτων να βελτιωθεί υπήρξε μία μέθοδος που έλεγε ότι ασκούμε πίεση για την καταβολή των κονδυλίων. Τι κάνατε, θέλετε καταρχήν βελτίωση. Και για να βελτιωθεί η καταγγελία, θυμάμαι ότι υπήρξε έκθεση πρωτοβουλίας του συναδέλφου Μουζότο, που δεν είναι πλέον βουλευτής, εδώ και πολύ καιρό. Και το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ακριβώς γι' αυτό το λόγο να παραπεμφθεί στο δικαστήριο η Γερμανία και η Ισπανία. Και χαίρομαι πολύ που είναι και η Γερμανία μέσα, αλλιώ θα νόμιζαν οι Ισπανοί ότι του καταδιώκω. Και ένα τέταρτο και τελευταίο. Στην έκθεση του Γενικού Διευθυντού για ε, τα περιφερειακά στη σελίδα 42, συγγνώμη, ε, ελπίζω να έχετε τα στοιχεία αυτά, λέει μια στατιστική εκεί για τις διορθώσεις του έτους 2008. Ο Ταμείο Συνοχής, Διαρθρωτικό κτλ κοινωνικό. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που δεν εκπροσωπούνται πουθενά. Όταν πρόκειται για νέα κράτη-μέλη το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν παλιά ε, κράτη όπως η Ιρλανδία που έχουν πάρει πολλά χρήματα και δεν αναφέρονται εδώ. Υπάρχει κάποιο παράρτημα, κάποια συμπλήρωση για αυτή τη σελίδα και από άλλες χώρες που δεν εμφανίζονται εδώ ή δεν ήταν στις προθέσεις σας, δεν το ψάξατε αυτό, δεν ξέρω. Θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περίπτωση της Ιρλανδίας, γιατί μέχρι το 2003 η Ιρλανδία αντλούσε πάρα πολλά κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Στην έκθεση του Γενικού Διευθυντού για τα κοινωνικά θέματα δεν έχουμε αποθεματικό για το σύστημα ελέγχου στη Βουλγαρία. Για ποιο λόγο. Δεν έχει καν εγκριθεί το σύστημα αυτό του ελέγχου. Δεν υπάρχει αποθεματικό επειδή δεν εγκρίθηκε. Για ποιο λόγο. Και πότε ε, θα έχουμε την έγκριση, την επικύρωση για να μπορούν να ξεκινήσουν και οι πληρωμές. Αυτά τα λίγο. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων από τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στην περίπτωση αυτή το είδος των στοιχείων που αναλύουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, οι λογιστικοί μηχανισμοί δηλαδή ελέγχου και ελεκτικό συνέδριο, είναι διαφορετικά από τα στοιχεία που αναλύουν οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές και νομισματικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το γνωρίζω το πρόβλημα αυτό, το έχω υπόψη μου για ορισμένα κράτη-μέλη και τα στατιστικά του στοιχεία. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή είναι διαφορετικά στοιχεία στατιστικά. Στην περιφερειακή πολιτική εργαζόμαστε με συναλλαγές, με πληρωμές, με δαπάνες είναι διαφορετικά από τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουν οι κατατόπους εθνικές υπηρεσίες ε, των κρατών μελών. Το αντικείμενο λοιπόν του ενδιαφέροντος μας είναι διαφορετικό από το οικονομικό και το νομισματικό. Είναι άλλη προσέγγιση. Και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουμε ε, σφάλματα και αμφιβολίες. Δεν έχουμε λόγο να αμφισβητούμε την αξιοπιστία των ε, στατιστικών στοιχείων που παρέχουν τα κράτη-μέλη οι λογιστικοί έλεγχοι γίνονται και εξυπηρετούν ακριβώς αυτόν τον σκοπό, να εντοπιστούν τα σφάλματα. Και όταν βρίσκουμε κάποια σφάλματα, τα διορθώνουμε. Είτε εμείς, είτε τα κράτη-μέλη. Μπορεί και η Επιτροπή να κάνει οικονομική διόρθωση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για το άλλο που ρωτήσατε. Εάν σε κάποιες περιπτώσεις Υπάρχουν εσφάλματα που επιμένουν. Αν έχουμε κανένα μηχανισμό, έτσι πώς να το πω, περικοπών ε, στη χρηματοδότηση των κρατών μελών αυτών. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε δύο περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας που αναφέρατε κι εσείς. Υπάρχει ένας μηχανισμός προοδευτικής ε, πάυσης, phasing out. Δηλαδή, οι δύο δικαιούχοι σιγά σιγά θα παίρνουν λιγότερα χρήματα μέχρι το 2010, αν δεν απατώ, με τα τέλη του 2010. Μιλώ για την ανάληψη υποχρεώσεων. Για την Ελλάδα δεν γνωρίζω τι με ρωτάτε. Uh, Θα πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό, να κοιτάξουμε γιατί λείπει η Ιρλανδική περίπτωση. Α, για τη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία έχουμε ακόμα πρόβλημα συμμόρφωσης και ε, εκτίμησης. Πολλά από τα προγράμματα που ε, ελέγξαμε και σε πολλές περιπτώσεις Ε, στοιχεία που μας έχουν δώσει οι βουλγαρικές αρχές τα έχουμε απορρίψει. Στο μεταξύ, άλλαξε η κυβέρνηση, ανέλαβε νέα. Είμαστε σε στενή επαφή με τη νέα κυβέρνηση και ε, φαίνεται ότι έχουν γίνει μεγάλες διοικητικές και ε, οργανωτικές αλλαγές και σύμφωνα με τόσο έχω υπόψη μου και τα, τις εκτιμήσεις δικές μου, οι νέες προσπάθειες που γίνονται από τη νέα κυβέρνηση είναι πραγματικά ελπιδοφόρες και τονίζεται η ανάγκη να υπάρχουν καλοί ε, μηχανισμοί ελέγχου της διαχείρισης. Πιστεύουμε δε ότι οι προσπάθειες αυτές αξίζουν υποστήριξη των υπηρεσιών μας και θα τις υποστηρίξουμε για να έχουν θετικά αποτελέσματα τους επόμενους μήνες. Βεβαίως, όλα αυτά είναι μάλλον μια εντύπωση που έχω εγώ παρά ε, ακράδαντη πεποίθηση. Ευχαριστώ. Θέλετε να παρέμβετε, κύριε Σπίτλα. Για την πρώτη ερώτηση. Για τη μήνυ δήλωση αξιοπιστίας. Θα ήθελα να σας πω ότι ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη και έδωσε σαφές αποτέλεσμα. Δηλαδή, ότι έχουμε νέους κανόνες για τη νέα προγραμματική περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών Βέβαια, ξέρετε ότι κάθε μεθολογία έχει τα ωριά της. Δεν μπορούμε να πούμε ότι βρήκαμε την πανάκια της μεθόδου και φτάσαμε στον τελικό μας στόχο. Ήταν ενδιαφέρον το εγχείρημα. Μη πείτε το τεστ, αλλά μας δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Θα ήταν όμως πρόωρο αυτή τη στιγμή να εξάγουμε συμπεράσματα για τη διαδικασία αυτή. Για την Ελλάδα, τώρα, το ελεκτικό συνέδριο στην πιο πρόσφατη του μελέτη, στη, στη, στο λογιστικό έλεγχο που έκανε, δεν βρήκε σφάλματα για την Ελλάδα. Μπορώ να σας πω ότι ήταν και από τα καλύτερα κράτη-μέλη στις επιδόσεις της η Ελλάδα στον τομέα αυτό. Για τη Βουλγαρία, στην περίοδο 2000-2006, η Βουλγαρία δεν πήρε τίποτα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν τα στοιχεία στη δήλωση του Γενικού Διευθυντή. Για τη νέα περίοδο δεν έχουμε τη δήλωση αξιοπιστίας. Επαναλαμβάνω, δεν έχει πάρει χρήματα από εκεί η Βουλγαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ω Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ζούμε μια σχιζοφρενική κατάσταση. Διότι εμεί ε, έχουμε ευθύνη να κοιτάμε πώς εκτελείται ο προϋπολογισμός, στα κονδύλια των φορολογουμένων. Μιλάμε για στατιστικά στοιχεία, για ε, δείκτες, για σφάλματα, πράγματα που συγκινούν τους δημοσιονομικούς ελεγκτές και τους συλλογιστές, αλλά θα πρέπει να δείχνουμε και κάποια ευθύνη. Όλοι εδώ γνωρίζουμε ότι στα θέματα τη εκτέλεση του προπολογισμού έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα κράτη-μέλη, τα οποία όμως θα πρέπει να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα πρέπει επίση να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώνουμε την κατάσταση. Εγώ είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένο και καθόλου δεν με ικανοποιεί ο τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται ε, σήμερα τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Επίσης είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την κατάσταση που επικρατεί στα γερμανικά ομόσπονδα κρατήδια των οποίων οι τοπικοί πρωθυπουργοί θέλουν να παίξουν και μεγάλο ρόλο στο μέλλον. Θα πρέπει να συζητήσουμε ε, όμως πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα τους φέρουμε ενώπιον των ευθυνών τους όλους αυτούς. Ας πούμε, έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση της διοίκησης των διαρθρωτικών ταμείων. Σα ρωτώ, για την πρώιμη φάση τη προγραμματική περίοδου 2000 με 2006, πόσα είναι τα κράτη-μέλη που δεν σας έχουν στείλει στοιχεία, που έχουμε ακόμα ελλείψεις στην καταγραφή της κατάστασης. Θα πρέπει να συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε ποιο φέρει ευθύνη γιατί. Τι έχει παραμεριθεί μέχρι τώρα. Τι θα αφήσετε στους ε, Αντικαταστάτε σα του διαδόχου Σα τι πρέπει να γίνει στο μέλλον για να μειωθούν τα σφάλματα και να ληφθεί υπόψη η ευθύνη των κρατών μελών με τρόπο που αρμόζει στο κάθε κράτος μέλος. Well, as I have already mentioned... Όπως είπα ήδη, η Κομισιόν έκανε διαβήματα και πήρε και πρωτοβουλίες στο πρόγραμμα δράσης ε, για να δώσει καλύτερες πληροφορίες στις κυβερνήσεις για τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν για τα διορθωτικά ταμεία. Ήδη είπα ότι η Κομισιόν δίνει διαφόρων ειδών πληροφορίες και προσφέρει κατάρτιση σε στελέχη που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των κονδυλίων των διαφορετικών ταμείων και έμεσα και ως προς τους δικαιούχους με δημοσιεύματα, με ηλεκτρονική διοχέτευση πληροφοριών Ένα από τα μείζωνα βήματα ήταν ένα σύνολο νέων κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με τις ε, ετήσιες συνόψεις που μας δίνουν με, τις οποίες, με τις οποίες μας δίνουν πληροφορίες οι κυβερνήσεις ως προς το τι προσπάθησε έκανε να βελτιωθεί η κατάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι ετήσιες συνόψεις επιβεβαιώνουν το ότι οι κυβερνήσεις όντως χρησιμοποιούν αυτές τις επιπλέον πληροφορίες της Κομισιόν. Βέβαια υπάρχουν και διαφορές από χώρα σε χώρα. Φυσιολογικό αυτό. Μερικές συνόψεις είναι πάρα πολύ καλές, μερικές είναι λιγότερο καλές. Η Κομισιόν θα συμπληρώσει το πρόγραμμα δράσης μέχρι το τέλος του χρόνου και θα σας τα αναφέρουμε αυτά το Φεβρουάριο. Φυσικά τα αποτελέσματα ως προς τα συγκεκριμένα νούμερα ή την επίπτωση αυτά θα τα έχουμε το 2010. οι δαπάνε που θα έχουν μελετήσει τότε, που θα έχουν, τις έχουν μελετήσει το Ελεκτικό Συνέδριο και ο Κομισιόν, αποκλειστικά θα είναι υπό, τις, υπό τη νέα προοπτική, με τη νέα μέθοδο διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζεται τώρα. Κύριε Πίπερτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ε, προς τον κύριο Σπίτλα είχε την καλοσύνη να μας πει ότι αν αποσυνδέσουμε από το κοινωνικό ταμείο, τα διαρθρωτικά ταμεία, λέει, θα πάνε όλα καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει το αντίστο. Αν θεωρήσουμε την κοινωνική πολιτική ως ξεχωριστό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό σημαίνει τεράστια αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μηχανισμούς ελεγκτικούς τεράστιους που δεν υπάρχουν και θα πρέπει να τους δημιουργήσουμε και δεν νομίζω η πλειονότητα των βουλευτών να βλέπει τα πράγματα όπως ο κύριος Σπίτλα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να κάνω ερώτηση στον κύριο Τσανέσκη. Έχουμε αυτό το 11% που είπαμε που κατανέμεται διαφορετικά στα κράτη-μέλη και στους ελέγχους των προηγουμένων ετών, για να μην πω δεκαετιών, έχουμε κατασυρωή κράτη που κάνουν επανειλημμένα κάτι λάθος και κατ' επανάληψη. Και ρωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκεφτεί ποτέ να κάνουμε διμερείς μηχανισμούς ελέγχου. Δηλαδή, η Ευρώπη και ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Διμερείς, επαναλαμβάνω, ελεκτικούς μηχανισμούς και παρακολούθησης, διότι δεν επιτρέπεται ολόκληρη Ευρώπη, 27 κράτη-μέλη, να υφίστανται τις συνέπειες ορισμένων που έχουν κακή συμπεριφορά κατά επανάληψη. Γιατί να το υφιστάμεθα όλοι αυτό. Το έχετε σκεφτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι στιγμής δεν ε, ελήφθησαν νομικά μέτρα από την Κομισιόν για διαφορετική μεταχείριση των κρατών. Ωστόσο, συζητάμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2013. Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις όπου Αφενός έχω μια διαφορετική προσέγγιση κατά κράτος, όπου ένα κριτήριο θα μπορούσε να είναι η ορθότητα των ελέγχων στο παρελθόν. Ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνη, ας πούμε, με τις χώρες που έχουν καλή επίδοση. όπου θα είμαστε λιγότερο σκληροί. και δίνουμε περισσότερη ευελιξία στο κράτος μέλος αμείβοντας την καλή συμπεριφορά. Από την άλλη μεριά διαφοροποιούμε τις μεθόδους επειδή η κατάσταση είναι διαφορετική. Αν συγκρίνουμε με το μέγεθος της διοίκησης και το μέγεθος των κονδυλίων κατά χώρα. Έχουμε χώρες, μεγάλες χώρες με λίγα κονδύλια για την πολιτική συνοχή δεν είναι σημαντικό το συνολικό ποσό και έχουμε μικρές χώρες, μικρή διοίκηση δηλαδή με μεγάλη ροή ε, κονδυλίων συνοχής. Δύο παράμετροι λοιπόν. Το μέγεθος της διοίκησης, το μέγεθος της χώρας ουσιαστικά, και το μέγεθος, το ύψος των κονδυλίων. Προκειμένου να έχουμε διαφορετικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Το συζητάμε ακόμη. Αυτό θα οριστικοποιηθεί το 2011. και. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία μικρή ερώτηση. Ο Επίτροπος Σεμέσκι πιστεύει ότι το 11% οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλματα και όχι σε απάτη. Ερώτημα. Το αν είναι λάθος ή απάτη εξετάται από την πρόθεση. Λάθος διαπράττουμε όταν δεν έχουμε καλή πληροφόρηση. Αν όμως πρόκειται για ένα λάθος που έγινε εν επιγνώση, είναι απάτη. Πού στηρίζεστε για να λέτε ότι πιστεύετε ότι δεν είναι απάτη. Στηρίζεται μόνο σε υπολογισμούς των κρατών μελών και το ηλεκτρικό συνέδριο τι λέει. Δεν υπάρχει ένα σκιώδες νούμερο όπου να μην ξέρουμε πρόκειται για λάθος ή για καθ' αυτό απάτη. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω, αν μου επιτρέπετε, ότι εμείς πιστεύουμε τα ευρήματα και το πόρισμα του ελεκτικού συναδρίου, όπου λέει ότι δεν ε, εμφανίστηκαν σφάλματα. Το σημειώνουμε με ικανοποίηση. Αν δούμε όμως τι είδους σφάλματα ανοιχνεύονται, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ακριβώς λόγω αυτού του ειδικού τύπου σφαλμάτων δεν υπάρχει πρόθεση που κρύβεται από πίσω, δηλαδή πρόθεση απάτης. Παράδειγμα. Στην περίπτωση σφαλμάτων σε προκήρυξη δημοσίων έργων ή όταν ε, προτείνονται κάποιες δαπάνες μη επιλέξιμες αυτό εύκολα φαίνεται ότι δεν ήταν ισχυμένο σφάλμα, δεν είναι απάτη αυτό. Αλλά νομίζω μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα το ελεκτικό συνέδριο γιατί δεν το κατατάσσουν σε, στην απάτη αυτό το φαινόμενο. <clears throat> Ο κύριος Όλμπριχτ. Ε, πρόεδρε, εάν ε, μου επιτρέπετε, θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στη διαδικασία της απαλλαγής και ιδιαίτερα για το 2008 είναι η ε, ανάλυση που λέει τι συνέβη ως αλλαγή από το 2006 και μετά, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι είχαμε άλλη διαδικασία στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και άλλα μέσα. Και μετά αποφασίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα αλλάξουμε. Παράδειγμα, να βγάλουμε την ανάπτυξη της πέθρου από την πολιτική συνοχής. Ή άλλο παράδειγμα, να αλλάξουμε ε, τον τρόπο χρηματοδότησης, να αλλάξουμε το σύστημα και να βάλουμε και για το Ταμείο Συνοχής τον κανόνα νη συν 2. Αυτό είναι πολύ σοβαρή αλλαγή και βεβαίως το θέμα δεν είναι του παρόντος, αλλά θα πρέπει να δούμε εάν έγινε αυτή η ποιοτική αλλαγή όταν αλλάξαμε τη μέθοδο. Μετά το 2006, αυτό είναι το ζήτημα. Όταν συζητήσαμε το περίφημο 100% το... Ελπίζω να μην είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη η συζήτηση για την πολιτική συνοχή σε αυτή καθ' αυτή. Να μην προσπαθούμε δηλαδή να αποδείξουμε ότι εξορισμό η πολιτική συνοχή προσφέρεται για απάτες και για σφάλματα. Καλύτερα να το αποφύγουμε. Αυτό θα πούν ορισμένοι. Δηλαδή, ορισμένοι θα πούνε α καταργήσουμε ολόκληρη την πολιτική αν δίνει έδαφο για σφάλματα και απάτε. Δεν είναι του παρόντο αυτή η συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δημόσια έργα, τι δημόσιε προμήθειες. δούμε το μεγάλο ποσοστό του 11% ε, συνδέεται άμεσα με δημόσιες προμήθειες. Τι τρέχει λοιπόν. Ε, μήπως υπάρχει κανένα ζήτημα επιλεξιμότητας. Άλλες αρχές έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιλεξιμότητα των ε, έργων από τις εθνικές διατάξεις. Αυτό είναι το θέμα. Πώς το αντιλαμβάνονται τα κρατη στους διαγωνισμούς για τις δημόσιες προμήθειες είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό για όλη την Ένωση. Εξού και η ε, πολιτική συνοχής που κατέδειξε το πρόβλημα. Δεν φταίει λοιπόν η πολιτική συνοχή. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στις ευρωκηρύξεις των δημοσίων έργων και ίσως και αυτό θα πρέπει να μας ε, προβληματίσει. Τι τρέχει με την επιλεξιμότητα και πώς γίνονται τα έργα. Αυτό είναι το ζήτημα. Πού είναι τα σφάλματα και τα προβλήματα στα δημόσια έργα. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναλύσουμε στο μέλλον. Μήπως πρέπει να εναρμονίσουμε περισσότερο το πρόγραμμα. Γιατί μόλις τώρα το φτιάξαμε. Μήπως στο μέλλον χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση. Οι κανόνες για την επιλεξιμότητα στην ίδια επένδυση, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικοί οι κανόνες, επαναλαμβάνω, από χώρα σε χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα πρέπει να πούμε στην ουσία του θέματος και να πούμε ότι χάρη στην πολιτική συνοχή καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς προκυρήσουν τα δημόσια έργα στην κάθε χώρα. Ευχαριστώ. Uh, <clears throat> Uh, Νομίζω ότι επί της αρχής συμφωνώ με την παρατήρηση που έκανε ο αξιότιμος Ευρωβουλευτής. Υπάρχει μια σειρά από σφάλματα τα οποία θα πρέπει να αποδοθούν στη στη διαφορετική χρήση των στοιχείων επιλεξιμότητας. Αν ο αντικειμενικός στόχος λοιπόν είναι να μειώσουμε τον αριθμό των λαθών, θα πρέπει να δούμε τι κανόνες ε, για την επιλεξιμότητα χρησιμοποιούνται και τι γίνεται με αυτούς που εφαρμόζονται για τη συνοχή. Μπορεί να είναι δεκτό από όλες τις πλευρές. Μπορεί να υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν διαφορετικά συστήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο για τους λόγους και μόνο της ε, ε, πολιτικής συνοχής νομίζω ότι είναι λογικό το επιχείρημα. Ευχαριστώ κύριο Σκάλφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση για τον Επίτροπο Σαμέτσκι. Είναι η υπεύθυνο για ένα χρονικό διάστημα για το οποίο δεν ήταν επίτροπος ε, λόγω των καταστάσεων. Και είναι και υπεύθυνο για μια στρατηγική τη οποία τα αποτελέσματα θα φανούν στην επόμενη θητεία της Επιτροπής. Ε, έχω μία ερώτηση. Έχουν ληφθεί πολλά μέτρα, έχουν υπάρξει βελτιώσεις το 2008, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για την απαλλαγή του 2008. Θα μπορούσατε να πείτε, κύριε Επίτροπε, ότι το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της προκειμένου τα ευρωπαϊκά κονδύλια να δαπονεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατά την άποψή σας, ε, τι γίνεται με τα διαρθρωτικά ταμεία, διότι εξ όσων γνωρίζω εγώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε το ίδιο ποσοστό σφαλμάτων και λήφθησαν ανάλογα μέτρα τα οποία οδήγησαν σε ανάλογα αποτελέσματα. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με τις μελλοντικέ ακροάσεις ε, των υποψηφίων επιτρόπων. Θεωρείτε ότι ο διάδοχός σας θα μπορέσει να αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις ε, για τα ποσοστά των σφαλμάτων και τα προγράμματα για τα οποία υπάρχουν παρατυπίες. Και μία τελευταία ερώτηση για την εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου το ελεκτικό συνέδριο μπορεί να εμβαθύνει περισσότερο όταν αναλύει το κατά πόσο χρησιμοποιούνται σωστά τα ευρωπαϊκά ταμεία. Για το πρώτο θέμα, σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ό,τι μπορούσε για να βελτιωθεί η κατάσταση το 2008. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν μια κάποια αδράνεια που οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμα το 2008 δεν είχαμε εφαρμόσει κάτι για τις νέες προοπτικές. Αυτές ε, που διαπιστώσαμε ήταν οι δαπάνες από το περίοδο 2000-2006 όπου είχαμε διαφορετικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Παραδόξως η σταθερότητα στα ποσοστά επιβεβαιώνει ότι τα θετικά αποτελέσματα θα παρατηρηθούν μόνο σε σχέση με τις δαπάνες λόγω των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Για το δεύτερο ερώτημα τώρα, για το αν αυτός που θα με διαδεχτεί θα μπορέσει να αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις. Αυτό θα το αποφασίσει αυτός βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα ήταν παρακινδυνευμένο να αναλάβει κάποιος ε, μετρήσιμες δεσμεύσεις, διότι ακόμα δεν έχουμε δει τι γίνεται στην πράξη και τι αποτελέσματα έχει. Νομίζω ότι το 2010 θα μπορούμε να πούμε ότι επειδή Το μερίδιο των δαπανών από τις νέες προοπτικές θα είναι περίπου 100% νομίζω το 2010. Όταν λοιπόν τότε έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα, ο νέος επίτροπος και οι υπηρεσίες του θα μπορέσουν να συζητήσουν σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό για να κάνουμε τις τελικές βελτιώσεις στο σύστημα. Επειδή όμως ακόμα δεν έχουμε τα πρώτα στοιχεία της συνολικής αλλαγής του συστήματος, θα ήταν παρακινδυνευμένο από πλευράς του. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε για ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω. Ευχαριστώ. Στο τέλος θα δώσω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε δύο-τρεις παρεμβάσεις ακόμα. Ο κύριος Γκάρικα Πογέδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Ο ένας από τους επιτρόπους της εξηγήσει του μας είπε ότι κάποιος δημοσιογράφος είχε πάρει κάποια λανθασμένα στοιχεία και δημιούργησε μια συγκεχημένη εντύπωση για το πώς έχει η κατάσταση για την εκτέλεση των ε, προϋπολογισμών των διαφθορετικών ταμείων. Αυτό που ζητάμε συνήθως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να μας δίνει τα στοιχεία όσο το δυνατόν πιο σαφώς και να έχουμε και όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Και όταν μιλάμε για δημοσιονομικές προοπτικές, συνήθως ε, μιλάμε για ε, καθαρή απώλεια κονδυλίων. Δεν είμαστε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και γι' αυτό λοιπόν δεν είμαστε υποχρεωμένοι να καταλαβαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, αλλά συνήθως όταν γίνονται διορθώσεις από ένα κράτος μέλος, υπάρχει δυνατότητα να γίνει ανακατανομή των κονδυλίων που κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δαπανήθηκαν σωστά και να πάνε σε άλλα κοινοτικά προγράμματα. Επομένω, η καθαρή απώλεια ποσών που μπορεί να έχουμε από τα διαθερωτικά ταμεία και από το Ταμείο Συνοχή θα πρέπει να συσχετίζονται με αυτά που υλοποιεί άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας δώσω εδώ το παράδειγμα της Ισπανίας, η οποία αναφέρθηκε επανειλημμένως. στο 60 δις ευρώ που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισπανία συγγνώμη, τα τελευταία χρόνια από το ε, ταμεία, διαρθρωτικά ταμεία και ε, το Ταμείο Συνοχής ε, δεν ξεπερνούν το 1%. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ελάχιστο ποσό, διότι δεν μιλάμε για απάτε, μιλάμε για δυσκολίε διοικητική φύσεω που ορισμένε φορέ ε, οδηγούν σε απώλεια κοινοτικών ε, κονδυλίων. Αλλά είμαστε στο 1%. Δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη που πρέπει να δει τι αποτελεσμάτα έχει η περιφερειακή πολιτική σε ένα κράτο μέλο. Αλλά η εκτέλεση ενό προπολογισμού 60 δι με όλα τα προβλήματα που έχει νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για τον τρόπο που μπορεί ένα κράτος μέλος να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί τα κονδύλια αυτά. Το σύνολο βέβαια μπορεί να είναι πολύ χειρότερο διότι το σύνολο του ποσού που διαχειρίζονται τα ταμεία μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που διαχειρίζονται άλλα κράτη-μέλη. Τώρα, στην παρούσα περίοδο προγραμματισμού από το 2007 και μετά, όπου είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό διορθώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση σαν αυτή που ήμασταν στο, και στο παρελθόν. Δεν έχουμε ένα σαφές πλαίσιο, δεν έχουμε τις καθαρές απώλειες από την αρχική περίοδο προγραμματισμού και ακόμα δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα. Πολλό δε μάλλον βεβαιασμένα συμπεράσματα. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν και από τους δύο επιτρόπους ε, και αυτούς και τους διαδόχους τους ε, που θα, τους, ε, που θα αναλάβουν καθήκοντα από το Φεβρουάριο να μας δίνουν πολύ πιο ενδελεχή στοιχεία για το τι γίνεται με την εκτέλεση και τις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις αυτή τη νέα περίοδο προγραμματισμού έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και να μην λαμβάνουμε βεβαιασμένε αποφάσει οι οποίε ορισμένε φορέ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρέγω. Μπορώ να σας δηλώσω ότι στο μέλλον θα σας δίνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των διορθώσεων με επιμερισμό κατά χώρα, κατά κονδύλι, ταμείο, για να μπορείτε να συγκρίνετε τη σχετική σημασία των διορθώσεων κατά χώρα. Πρόεδρος. Έχω και εγώ να κάνω μερικές ε, ερωτήσεις και σχόλια. Κύριε Επίτροπε, στην αρχή μας είπατε ότι να διασκεδαστεί η παρανόηση μεταξύ λάθος και δόλου ή απάτης. Η Επιτροπή μας έχει δικαίωμα να καταλάβει πού είναι τα λάθη και πού είναι ο δόλος. Και νομίζω όλοι στόχο μας έχουμε να μην ε, να ξεπεράσουμε την τυπολατρεία όπου, ε, που εμποδίζουν την αποτελεσματική χρήση των κοδηλιών όμως. Στόχος μας επίσης όλοι να έχουμε ανοχή μηδέν ως προς τις απάτες. Εγώ δεν είμαι τόσο πεπισμένος όσο εσείς ότι 2008 δεν υπήρξαν απάτες. Το αν δεν καταγράφηκαν θα πρέπει να ελέγξουν τα ελεγκτικά όργανα περισσότερο. Η όλα Φερρυπίν, κατά πόσο αυτοί οι δείκτες που θεωρούνται σοβαροί από το ελεγκτικό συνέδριο για τις δημόσιες προμήθειες, διορθωτικά προ, ε, προγράμματα, συνοχή, σοβαρές περιπτώσεις. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να έχουμε παρατυπίες, άλλες λιγότερες. να αναφέρετε την Απολία και την Καλαβρία. Εγώ δεν είμαι καθόλου πεπισμένο ότι είναι παρατυπίες και όχι απάτες. Γι' αυτό δεν το λέω ως πρόεδρος τη Επιτροπής, αλλά επειδή μας το λένε ένα σωρό έρευνας που το έχει κάνει η ειδική αστυνομία, φοροαστυνομία, δικαστές. Χρειάζεται να καταβάλουμε ακόμα περισσότερη προσπάθεια γιατί ο ελεκτικό συνέδριο έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά πρόσφατα με ένα σωρό δείκτες και τυπικών σφαλμάτων αλλά και σοβαρών παραβάσεων της νομοθεσίας. Και η ερώτησή μου είναι η εξή. Την έκαναν και άλλοι συνάδελφοι. Θα την κάνουμε και στους νέους επιτρόπους, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση μπορούμε νομικά να προβλέψουμε κυρώσεις κατά των κρατών που δεν συμμορφώνονται και που επαναλαμβάνουν το ίδιο. Γιατί είπατε το ίδιο πρόβλημα θα το συναντήσουμε το 2000, θα το αντιμετωπίσουμε το 2013. Ήδη από το 2006 είχαμε στοιχεία που μας τα δείχναν αυτά. Είχαμε ενδείξεις ότι υπάρχουν χώρες που συστηματικά παραβιάζουν διαδικασίες προκειμένου να δοθούν δημόσια κονδύλια. Και πέρα από τις νομικές κυρώσεις έχουμε και πολιτικές κυρώσεις. Γιατί εγώ θεωρώ άτοπο, απρεπές να υπάρχουν χώρες που συστηματικά τηρούν τους κανόνες και άλλες χώρες που τις ξέρουμε καλά και ακούσαμε ποιες είναι, πάνω κάτω ίδιες, προξενούν μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για τις άλλες χώρες της Ένωσης, κυρίως για τις χώρες που παίρνουν τα λεφτά, γιατί οι πολίτες αυτών των χωρών που παίρνουν τα λεφτά βρίσκονται πάντα στη μαύρη λίστα. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Ούτε για αυτούς τους πολίτες του, για την εικόνα της χώρας. Σας καλώ λοιπόν αυτό το τις αιτιάσεις μου και αυτό το αίτημά μου αν θέλετε να τα φέρετε στους νέους επιτρόπους μην ξανασυζητάμε το 2013 ότι υπάρχουν χώρες και περιφέρειες χωρών που είναι συνεχώς το μαύρο πρόβατο. Well, thank you for suggesting... Σας ευχαριστώ που μας προτείνετε να διαβάσουμε ε, τα μηνύματα αυτά στους αντικαταστάτες, στους ε, επιτρόπους που θα μας διαδεχτούν και βέβαια θα το κάνω κι εγώ. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, έχει βρει κανένα λόγο, ε, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα έτσι ώστε οι παρατυπίες ή τα σφάλματα που έχουν βρεθεί για το 2008 να χαρακτηριστούν απάτη. Κατά την άποψή μου και την γνώση μου, όταν υπάρχουν ε, ύποπτε περιπτώσεις διαβιβάζονται στην υπηρεσία της Όλαφ που είναι το αρμόδιο όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επαληθεύσει και να ελέγξει σε ποιο βαθμό αυτά συνιστούν ε, απάτη. Αυτές οι υποψίες είναι βάσιμες ή αβάσιμες δηλαδή. Από την παρελθούσα εμπειρία ε, φάνηκε ότι μόλις 0,11% του συνόλου των δαπανών του ετησίου προϋπολογισμού για τη συνοχή ε, θεωρήθηκαν ε, ύποπτη απάτη, ύποπτη και πάλι όχι επιβεβαιωμένη και αποδεδειγμένη, ύποπτη απάτη. Το ένα εκατοστό δηλαδή από το δίκτυ ε, σφαλμάτων. Και πάλι επαναλαμβάνω πρόκειται για υποψίες απάτης και όχι για επιβεβαιωμένες περιπτώσεις απάτης. Για τις νομικές κυρώσεις τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει τέτοιου είδους κυρώσεις κατά των κρατών μελών που επίμονα ε, έχουν κακές επιδόσεις ε, στον τομέα αυτό. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να φανταστούμε τέτοιου είδου κυρώσει, αλλά αυτέ θα πρέπει νομικό κανονισμό ή κανονισμού ή στι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ από το 2013 και μετά. Εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία σας, Πρόεδρε, ε, για την ανάγκη ε, άσκησης πίεσης στα κράτη-μέλη εκείνα που έχουν τις πιο κακές επιδόσεις και μία από τις παρακαταθήκες μου για το μέλλον θα ήταν να οργανωθεί υψηλού επίπεδο πολιτική συζήτηση σε υψηλό επίπεδο, ας πούμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων άπαξ του έτους, ε, σχετικά με τις επιδόσεις και τις, ε, ε, την κανονικότητα των δαπανών κτλ. Αν μη τι άλλο να υπάρχει μία πίεση μεταξύ των κρατών μελών, από τους ομολόγους τους όμως, αυτό και πάλι η πρόταση δική μου είναι, δεν είναι, η πρακτική που υιοθετείται ως τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ σε ευχαριστώ κύριο Σπίτλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα σύντομα να προσθέσω κάτι κι εγώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίε τη έχουν μηδενική ανοχή, όπως είπαμε, απέναντι στην απάτη. Δηλαδή, όλες οι περιπτώσεις που θεωρούμε ότι ενδεχομένω ε, τα σφάλματα παραπέμπουν σε απάτη, διαβιβάζονται στην Όλαφ, που είναι το αρμόδιο όργανο. Το είπε ήδη ο συναδελφό μου προηγουμένω. Και μάλιστα είπε και ε, ε, πόσα χρήματα είναι αυτά για τα οποία συζητούμε. Κάτι άλλο που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι πώς θα βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν έχουμε περιπτώσεις με υποψία απάτης. Αυτό ναι, είναι ένα ζήτημα πρακτικό προς συζήτηση. Ωστόσο θα πρέπει να σας πω ότι η ανοχή μας απέναντι στην απάτη είναι μηδενική. Αλλιώς θα διακυβεύαμε την ίδια την ουσία της πολιτικής συνοχής και της ε, πολιτικής. Επειδή δεν έχουμε χρόνο πια, πολύ σύντομα η Στάφη Άντριάσεν και μετά ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου που έχει μια ερώτηση από τους συνδέφους Κάλλη και Ζόντεργερ και στο τέλος ο συγητής Λιμπεράσκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι σε θέση να πούνε αν αυτό είναι λάθος ή απάτη. Διότι όλοι μιλάνε για την εγκληματική πρόθεση. Αυτό μπορεί να κριθεί μόνο από μία ποινική, ποινικού χαρακτήρα έρευνα, αστυνομία. Το αν είναι λάθος ή απάτη, για μένα η διάκριση είναι πολύ ασαφής είναι πολύ δύσκολο αυτά τα όργανα να το ορίσουν. Αλλά ξανάρθουμε σε αυτό που είπε το ηλεκτρικό συνέδριο. Το να ζητάει κανείς κονδύλια όταν δεν είναι επιλέξιμος είναι κακή χρήση, κατάχρηση καλύτερα των χρημάτων του φορολογούμενου. Επίσης, ευχαριστώ την προσοχή σας ότι το ηλεκτρικό συνέδριο λέει όταν λύγει η περίοδος εφαρμογής ενός προγράμματος αυξάνει ο κίνδυνος και ρωτώ την Κομισιόν έχει σχέση αυτό με τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζουμε τον προπολογισμό ή όχι. Τρίτον, σε σχέση με αυτά που είπε ο Επίτροπος Σενέκη στις απαντήσεις του στην αρχή, να προτείνουμε εμεί να αλλάξουν οι δημοσιονομικοί κανονισμοί ώστε να μπορούν να διακοπούν οι πληρωμές αν θεωρηθεί ότι έγινε κατάχρηση των κονδυλίων. Απάντηση σύντομα. Vuole rispondere? In attesa. In attesa do la parola al rappresentante della Corte dei Conti. Prego. Εν αναμονή να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την απάτη. Ένα σύστημα που δεν αποδίδει ε, τίνει προς απάτη, όχι μόνο προς λάθη. Μικρά τυπικά λάθη που δεν είναι καν ποσοστοποιήσιμα μπορεί να οδηγήσουν σε μεθέσεις που μπορεί να συμβεί απάτη. Πρέπει να δημόσιες προμήθειες μπορεί να γίνει ένα σχέδιο να μην υπάρχουν υποψήφοι για ένα κείμενο, να μην υπάρχουν έγγραφα ότι έγινε ανοιχτή η διαδικασία με την ανακοίνωση του διαγωνισμού κλπ. Αν δεχτούμε αυτά τα λάθη και δεν τα διορθώσουμε αμέσω, έχουμε ένα σύστημα που θα επιτρέψει να περάσει η απάτη. Είχαμε περιπτώσει αυτά τα μικρά τυπικά λάθη συναθρίζονται και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να, να, να πούμε ότι έγινε σωστά η δημόσια προμήθεια. Είναι σωστά, κύριε Ανδριάσεν. Δεν ξέρουμε αν είναι αμέλεια ή απάτη. Φυσικά ο δικαστής, ε, ο ανακριτής θα το κρίνει αυτό. Υπάρχουν όμως συστήματα που δεν λειτουργούν και τα συστήματα αυτά τίνουν προς απάτη. Ερωτήθη αν το ηλεκτρικό συνέδριο μπορεί να πάει πιο περισσότερο σε βάθος αναλύοντας την, την, το σύνομο των πράξεων. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το μοντέλο διασφάλισης στοιχίζει πολύ. Μπορεί να χρειάζονται τρει ειδικέ εκθέσει, παραδείγματο χάρη, για μία συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή σα ενδιαφέρει πώ δαπανώνουν τα χρήματα. Το θέμα αυτό πρέπει να το συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά, αν θέλετε, στο μέλλον. Πρόεδρο, και δύο λεπτά για τον εισηγητή μα, τον κύριο Λιμπεράτσκι, και κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή συζήτηση μας δείχνει ότι ακόμα δεν βρισκόμαστε κοντά σε μια καλή συζήτηση. Παραδείγματος χάρη σφάλμα, απάτη. Για τα σφάλματα είναι κάπως σαφής η κατάσταση. Για την απάτη τα πράγματα περιπλέκονται. Αλλά δεν, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ε, παραλύσει το σύστημα των υπέρ των δικαιούχων. Τον ελέγχουν βέβαια του λογαριασμού μετά από 10 χρόνια. Και το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρεται μέχρι το έτος 2000, 2006. Στο τέλος του 2008 ο Επίτροπος Αμέσκη μας λέει δεν αναφερθήκαμε στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013. Η Κομισιόν είναι ανήμπορη μπροστά σε αυτό. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό. Μια ερώτηση προς τους επιτρόπους δεν λέμε καλύτερα ποιες είναι οι χώρες αυτές. Πριν ο Επίτροπος μας είπε ότι δεν πληροφορήθηκε ακριβώς σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού των σφαλμάτων εκ μέρους του ελεκτικού συνεδρίου. Ταυτόχρονα θέλει να συνεχίσει με τα mini για το 2007-2013. Το ελεκτικό συνέδριο επ' αυτού τι λέει. Τι λέει για τη θέση αυτή της Κομισιόν. Δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο, αλλά κάπου διαβάσαμε ότι υπάρχουν όλο και λιγότερες αποφάσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Αυτές οι διορθώσεις συχνά θεωρούνται από τα κράτη-μέλη ως κύρωση. Πώς είναι δυνατόν να ασκήσουμε πίεση σε μια χώρα αν αυτές οι οικονομικές διορθώσεις χρησιμοποιούνται όλο και πιο λίγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί πολλές ώρες. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε χρόνο. Τα ερωτήματα του εισηγητή θα διερευνηθούν σε επόμενη συνάντηση. Ευχαριστούμε τους Επιτρόπους για την γόνιμη αυτή συζήτηση. Και τώρα πρέπει να περάσουμε στο σημείο 5. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Καλώς ορίσατε στον πρόεδρο Μεστάντ. Του δίνω μέσα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Να λάβω το λόγο και πάλι στην Επιτροπή σας, διότι όντως παρόλο που δεν προβλέπει τίποτα η συνθήκη σχετικά, εγώ θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό ο πρόεδρος ενό Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου να κληθεί ή να καλείται καλύτερα να απαντά στι ερωτήσεις των ε, προσώπων των Ευρωπαίων πολιτών. Σα έχω διαβιβάσει και επιστολή άλλωστε για τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις των διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια. Θα είδατε ότι σχεδόν το σύνολο των συστάσεων που εξαρτώνται από εμά έχουν τεθεί σε ισχύ. Έχετε κάνει βέβαια και πολλές συστάσεις που δεν είναι μόνο αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στην έκθεση για το 2006, ο κύριο Οντί επέμεινε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έχει μια τραπεζική υποπτία. Αμέσως εγώ δήλωσα την προθυμία της τράπεζας να υπόκειται σε ένα τέτοιο έλεγχο, αλλά είναι αυτονόητο ότι αυτό δεν εξαρτάται από μας. Η πιο αυτονόητη λύση που σκεφτήκαμε όλοι θα ήταν να ε, υποκληθούμε στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί από τη συνθήκη του Μαστρίχτ αυτό προβλέπεται. Αλλά για να τεθεί σε ισχύ χρειάζεται ομοφωνία των κρατών μελών και παρά τις επανειλημμένες απόπειρε φαίνεται ότι δεν υπάρχει ομοφωνία των κρατών μελών για να αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την εποπτεία της Τράπεζας Επενδύσεων. Εν παρόδο θα σας ε, πω ότι θα έχετε την ευκαιρία να επανέλθετε σε αυτό γιατί το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ σήμερα συζητήσαμε μια πρόταση ε, για την ε, τραπεζική εποπτεία, πρόταση η οποία έρχεται να τροποποιήσει τη σημερινή ΣΕΠΣ σε μια ευρωπαϊκή αρχή για τις τράπεζες και το κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο δεν προβλέπει τίποτα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΜΕΝ, αλλά αν μου επιτρέπετε, σας προτείνω να επανέλθετε, αν θέλετε, στο θέμα αυτό και να προτείνετε μεταξύ των νέων αποστολών αυτής της νέας αρχής να είναι και ένα είδος εποπτείας επί της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων. Οπότε σήμερα εμείς επαναλαμβάνουμε και πάλι την προθυμία μας να ελεγχόμαστε. Στο μεταξύ, τέθη σε ισχύ η συνθήκη της Σαβώνας που προβλέπει ενίσχυση της Επιτροπής Επαλήθευσης, Comité de Verification, που όπως γνωρίζετε αναφέρει άμεσα ε, στους διευθυντές ε, και ε, θα διπλασιαστούν τα μέλη από τρία θα γίνουν έξι και μπορούμε επίσης να διορίσουμε παρατηρητές, όχι η τράπεζα αλλά η Διευθυντική Επιτροπή. Και θα προτείνουμε στη Διευθύνουσα Επιτροπή ε, και στη νέα επιτροπή μάλλον ε, της επαλήθευσης που θα είναι ισχυμένη να έχουμε και εμπειρογνώμονες της τραπεζικής εποπτείας. Αυτή η επιτροπή θα έχει όχι απλώς τους ε, λογαριασμούς και την κανονικότητα των οικονομικών συναλλαγών, αλλά και τα πόσο συνάδουν όλα αυτά με τις βέλτιστες πρακτικές. Τις τραπεζικές πάντα. Λοιπόν, αναμένοντας πιο ο, ριζικές αν θέλετε σχέσεις και λύσεις ε, σας προτείνουμε αυτό τώρα για τη Βασιλεία 2 και πάλι δεν είμαστε υποχρεωμένοι αλλά εθελοντικά αποφασίσαμε να επιλέξουμε και να εφαρμόσουμε την πιο ε, προηγμένη φόρμουλα της Συμφωνίας Βασιλεία 2 για να γίνει αυτό Χρειάζομαστε συμβουλές και εποπτεία αρμοδίων και αρχών και προς το παρόν είναι η αρχή του Λουξεμβούργου που μας βοηθάει. Από φέτος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης είναι επιλέξιμη ως συνομιλητής της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη νομισματική πολιτική και αυτό μας υπέβαλε σε μια σειρά ε, απαιτήσεων αναφορών και πληροφόρησης ε, παρά τη έκτα ε, για να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο ρευστότητας. Και πρέπει να σας πω ότι όσοι ασχολήθηκαν με αυτό εξεπλάγησαν από τόσο προηγμένο είναι το σύστημα διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας που διαθέτουμε και πόσο σοφιστικέ. Συστάσεις λοιπόν του Κοινοβουλίου δίνουμε συνέχεια και θέλουμε να δοθεί συνέχεια αλλά δεν είναι απόλυτα στο χέρι μας αυτό. Κατά τα λοιπά, είναι σαφές ότι φέτος η βασική μας ανησυχία και μέλημα ήταν να απαντήσουμε ε, στην, ε, στο αίτημα των κρατών μελών να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της οικονομικής και νομισματικής κρίσης. Γι' αυτό αυξήσαμε πολύ τα δάνεια φέτος. Πριν από το 2007 και την κρίση δανείζαμε 45 δισεκατομμύρια στην Ένωση το χρόνο και φέτος 75 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 70 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ουσιαστική η αύξηση αυτή και κυρίως βασίζεται, όπως μας ζήτησαν οι μέτοχοί μας, κυρίως βασίζεται και κατευθύνεται σε τρεις κατευθύνσεις. Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ένα νέο είδος, με νέα φόρμουλα ε, δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παίρνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, με την προϋπόθεση ότι ε, χρησιμοποιούν τα κονδύλια αυτά για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων. Και έχουμε νέου είδους σύμβαση με πολύ πιο αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για διαφάνεια και για πραγματική χρηματοδότηση των μικρομεσαίων από τι τράπεζε. Δεύτερο κατεύθυνση προτεραιότητας είναι η κατευθυνση προτεραιότητα ειναι έργων για την καταπολέμηση της κλιματική αλλαγή και φέτο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ προγράμματα που άμεσα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου Μερικά στοιχεία θα σας δώσω συντομία, γιατί δεν είναι κοινοθέν που έχει πολλά λάθη σχετικά σήμερα. Το 2008, 2 δις, 2 ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φέτος θα είναι 2,5 δις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι πάνω από τη μισή χρηματοδότηση για την παροχή και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παραμένω στην ίδια κατεύθυνση κατά πολέμηση κλιματικής αλλαγής. Έχουμε ένα νέο μέσο, μια νέα διευκόλυνση που ονομάζεται ECTF για προγράμματα έρευνας για καθαρές τεχνολογίες μεταφορών, για κινητήρες καθαρούς, για κάψιμα πιο καθαρά, για να μειώνονται οι εκπομπές και κυρίως να μπορούν τα αυτοκίνητα να σέβονται τους νέους ε, κανόνες ε, για τα καυσαέρια που θα τεθούν σε ισχύ το 2015. Και ο τρίτος προσανατολισμός που μας τέθη από τους μετόχους μας είναι να κάνουμε φέτος μια ιδιαίτερη προσπάθεια επιταχύνοντας την εκταμίευση σε χώρες και περιφέρειες που επλήγησαν σοβαρότερα από την κρίση. Γι' αυτό φέτος λοιπόν Έχουμε δανείσει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν στις χώρες της Βαλτικής, στην Ουγγαρία ή τη Ρουμανία, για να αναφέρω απλώς και μόνο μερικές χώρες που ξέρετε ότι επλήγησαν ε, περισσότερο και πιο σκληρά. Άλλο στοιχείο επικαιρότητα, σας είπα, τέτοια ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και ε, σε παράρτημα συνάπτεται ένα πρωτόκολλο που τροποποιεί ε, το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έξι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις είναι αυτές. Πρώτον, τροποποίηση καλύτερα. Ε, ανάληψη περισσότερου κινδύνου, γιατί θεωρούν ε, φυσιολογικό να αναλαμβάνει τον κίνδυνο η τράπεζα. Μέχρι τώρα όταν έπρεπε να ανοιγόμαστε περισσότερο στον κίνδυνο από ότι μια εμπορική τράπεζα θα έπρεπε να έχουμε ειδική πρόβλεψη. Αυτό πλέον καταργείται. Δεν είναι απαραίτητο γιατί με βάση τη νέα συνθήκη θεωρείται η ανάληψη κινδύνου μια φυσιολογική αποστολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βεβαίως πάντα γίνεται αυτό με τρόπο πάρα πολύ ε, σόφρονα, δεν θα το ρηψοκινδυνεύσουμε κιόλα, αλλά έχουμε περισσότερη ευελιξία για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε με μεγαλύτερο κίνδυνο κάποια έργα, ιδιαίτερα κάποια ερευνητικά έργα και προ την ανάπτυξη. Δεύτερη τροποποίηση από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Στο εξή, τεχνική υποστήριξη που είχαμε μέχρι τώρα αναπτύξει πολύ περιορισμένα και πάντα σε άμεση σχέση με συγκεκριμένο δάνειο. Η τεχνική λοιπόν αυτή υποστήριξη πλέον γίνεται γραμμή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με βάση οδηγίες που θα εγκρίνουν η ε, Διευθύνουσα Επιτροπή της. Τρίτη τροποποίηση. Εις το εξή, χωρίς να χρειάζεται να εγκριθεί συνθήκη, θα μπορούμε να δημιουργούμε θυγατρικές, ε, εφόσον υπάρχει ομόφωνη ε, συμφωνία της Διευθύνουσης Επιτροπής. Τέσσερα, Τέταρτη τροποποίηση, αν αυτό χρειάζεται θα μπορούμε άμεσα να παίρνουμε μερίδια συμμετοχής σε επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν με τρόπο έμεσο, με ε, διαρθρωτικά ταμεία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, ανάληψης μεριδίων σας λέω ευθύ εξ αρχής ότι δεν θέλουμε καθόλου να αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ως ενδεχόμενο και σε έκτακτες περιστάσεις μπορεί αυτό να αποφανεί χρήσιμο, όπου θα θεωρούσε σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μερίδιο σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Πέμπτη τροποποίηση. Gearing ratio λέγεται, που είναι ο ε, λόγος ε, ανάμεσα στους ιδίους πόρους μας και στο σύνολο της δανειοδότησής μας. Ε, σύμφωνα με τη συνθήκη της Αβώνας, οι ίδιοι πόροι μας ορίζονται με τρόπο πιο ευρύ. Έτσι έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο χειρισμών. Και η έκτη τροποποίηση, το είπα προηγουμένω, ενισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα στο ρόλο τη Επιτροπή Επαλήθευση, αυξάνοντα τον αριθμό των μελών τη αφενό και αφετέρου ε, επιφορτίζοντα τον με την τον έλεγχο κατά πόσο εμείς έχουμε συμμόρφωση προς τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές. Αυτά. Το 2010 σίγουρα θα απασχολήσει πολλές επιτροπές του Κοινοβουλίου η συζήτηση για την αναθεώρηση των εξωτερικών μας εντολών. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ουσιαστικά και κανονικά δραστηριοποιείται στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 90% των ε, συναλλαγών μας είναι στο εσωτερικό της Ένωσης. Για να δράσουμε εκτός Ένωσης, αυτό ε, επιτρέπεται, αλλά πρέπει να έχουμε εντολή που μας τη δίνει είτε μια συνθήκη, είναι η Συμφωνία Κοτονού για τις χώρες ΑΚΕ, είτε απόφαση του Συμβουλίου που ορίζει και ένα πλαφόν, το μέγιστο ποσό που μπορούμε να δώσουμε ως δάνειο σε μια περιφέρεια, για ποιο είδους έργα και με ποιες προϋποθέσεις. Σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ασάφεια, διότι έχουμε πολλές εντολές διαφορετικές και ε, με τρόπο πολύ διαφορετικό φτιαγμένες. Μπορούμε σε μια περιοχή του κόσμου να δραστηριοποιηθούμε, κάπου αλλού όχι, ή σε ένα είδους έργο σε κάποια περιοχή, το ίδιο έργο αλλού όχι. Άλλες φορές η εντολή μας είναι αναπτυξιακού τύπου, άλλες φορές καθόλου, απλώς υποστήριξη ευρωπαϊκών συμφερόντων σε μια περιοχή του κόσμου. Με δύο λόγια, η αναθεώρηση των εξωτερικών εντολών προσφέρεται για διευκρίνηση και για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί μετά απόφαση του ΔΕΚ αυτές οι αποφάσεις για τις εξωτερικές εντολές δεν λαμβάνονται μόνο από το Συμβούλιο, είμαστε πλέον στη συναπόφαση με το Κοινοβούλιο. Και ένα τελευταίο, Πρόεδρε, δύο λόγια μόνο για την επιθυμία διαφάνειας και καταπολέμησης κάθε είδους ε, απάτης ή ε, διαφθοράς. Ε, σας είπα ότι έχουμε μηδενική ανοχή για την απάτη και για τη διαφθορά από τη στιγμή που ένα μέλος του προσωπικού έχει ε, αποχρώσει, ε, ενδείξεις ότι μπορεί κάπου να υπάρχει ε, απάτη ή διαφθορά που δραστηριοποιούμαστε εμείς, θα πρέπει αμέσως να το καταγγέλει και δυστυχώς αυτό συμβαίνει κατά καιρού. Έχουμε νέους κανόνες για να προστατεύουμε εκείνους που καταγγέλουν αυτά τα φαινόμενα και να αισθάνεται άνετο ο καθένας να αποκαλύπτει ε, μια διαφθορά ή μια απάτη, ακόμα και αν πρόκειται για το εσωτερικό. Οι λεγόμενοι whistleblowers, λοιπόν, εκείνοι που ε, αποκαλύπτουν αυτά τα θέματα, προστατεύονται και μάλιστα έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την OLAF, ε, την Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης. Τώρα, για τη χρηματοδότηση offshore το συζήτησαν οι 20. Ε, μάλλον για, για τα offshore ε, κέντρα ε, χρηματοπιστωτικά κέντρα, τα υπεράκτια. Ε, έχουμε τη στάση του G20. Βεβαίως υπήρχε από το παρελθόν απαγόρευση να χρηματοδοτούμε offshore φορείς στη μαύρη λίστα προφανώς διατηρείται αυτή η απαγόρευση, αλλά... Α, εκτός αν πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο, το οποίο βρίσκεται στην λόγω χώρα, έτσι, στην επικράτεια της χώρας, πάντα ελέγχουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με φοροδιαφυγή ή παράνομες πρακτικές. Λοιπόν, δεν χρηματοδοτούμε ε, εταιρείε που εδρεύουν σε ε, χώρε τη μαύρη λίστα. Αλλά κάναμε ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει και Θεά λίστα του ε, ΟΣΑ που λέγεται monitor jurisdiction, κάποιε δικαιοδοσίες υπό παρακολούθηση. Αν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε μια τέτοια εταιρεία, ζητούμε μετεγκατάσταση, να εγκατασταθεί αλλού, εκτός ε, της γκρίζα λίστης. Ε, για πρώτη φορά το εγκρίναμε αυτό, είμαστε ο πρώτος διεθνής οργανισμό και ελπίζουμε να μας ακολουθήσουν και οι άλλοι, έτσι ώστε να διατηρηθεί η πίεση αυτή. Τώρα, σε όλα μα τα νέα κείμενα συμβάσεων έχουμε μια διάταξη που προβλέπει ότι σε περίπτωση που η χώρα στην οποία εδρεύει η εταιρεία αυτή πέσει στον κρίζο κατάλογο, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, είναι ρευστά, τότε θα πρέπει ε, ε, μέσα σε ένα χρόνο να μετεκατασταθεί ή να εξοφλήσει το δάνειο της τραπέζης. Δηλαδή, εκεί πραγματικά πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε στην αιχμή του δόρατος της καταπολέμησης των καταχρήσεων αυτών των ε, υπεράκτιων χρηματοοικονομικών κέντρων. Για τη διαφάνεια, αν είχατε την περιέργεια να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, θα διαπιστώσετε ότι σήμερα έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες ε, από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Θα δείτε στον ιστότοπό μας, ας πούμε, και είμαστε το μόνο θεσμικό όργανο που το κάνει. Έχουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο για την επόμενη τριετία ε, με ποσά, σε κάθε κλάδο πόσα θα δαπανίσουμε, ποιες είναι οι πολιτικές δανειοδότησεις στους μεγάλους τομείς όπως είναι η ενέργεια, μεταφορές, για να ε, έρχεται στη συνέχεια να επαληθεύσετε εάν ανταποκρινόμαστε στις ε, πολιτικές. Στους κανόνες για το περιβάλλον και για την ε, κοινωνική πτυχή να παρακολουθείτε και σε περίπτωση που κάνουμε κάτι λάθος να μας το επισημάνετε. Επίσης να δείτε τον κατάλογο των έργων και των ε, σχεδίων που εξετάζουμε για να μπορέσετε να αντιδράσετε πριν το συζητήσει το Διοικητικό μας Συμβούλιο ε, επίση, θα βρείτε και πολλέ ΜΚΟ τα χρησιμοποιούν όλα αυτά. Θα βρείτε και τις εκθέσεις της ανεξάρτητης μονάδα μα για εκ των υστέρων αξιολόγηση. Και εκθέσει αυτέ καμιά φορά είναι επικριτικέ, διότι ό,τι έχουμε χρηματοδοτήσει στο παρελθόν δεν έχει στεφτεί με επιτυχία. Υπάρχουν και επικρίσει, οι οποίε είναι και δημόσιε στην ιστοσελίδα μα και οδηγούν και σε ε, ευρείε συζητήσει για να βελτιώνονται τα πράγματα στο μέλλον. Φροντίσαμε επίση να ε, εφαρμόσουμε τον κανονισμό 1367 του 2006 για τη σύμβαση άρχους για την πρόσβαση του κοινού δηλαδή στα έγγραφα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και αυτό άλλωστε είναι και αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης σε δύο γύρους μόλις ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος της δημόσιας διαβούλευσης και προσεχώς θα ε, αναθεωρήσουμε την πολιτική μας αυτή διαφάνειας και πρόσβαση στα έγγραφα. Αυτά πρόεδρε τα ολίγα και συντομία ως επισκόπηση των δραστηριοτήτων μας. Είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την σύνοψη και για τα πολύ σημαντικά στοιχεία που δώσατε στην Επιτροπή μας. Να δώσω το λόγο στον συγητή, τον κύριο Ντόιτς. <clears throat> Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριε Μάλστατ. Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ για την ε, έκθεση πολύ καλής ποιότητας που υποβάλλεται στην Επιτροπή μας και να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας εδώ. και για την προφορική παρουσίαση που κάνατε εδώ για να ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο σημαντικό για να ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι πολίτες. Η παρέμβασή μου θα εστιάσει σε τρία σημεία και από εκεί και πέρα περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα βελτιώσουν την έκθεσή μου. Θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τρία βασικά θέματα. όταν θα εξετάσουμε την έκθεση του 2008 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η τράπεζα δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια, επομένως θα πρέπει να δούμε τι πρόοδος επετεύχθη το 2008 πώς επηρεάστηκαν οι δραστηριότητες της τράπεζας από την χρηματοοικονομική κρίση κατά τη διάρκεια του 2008 και επίσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι προτάσεις που έγιναν κατά την τελευταία χρονιά υλοποιήθηκαν ή όχι κατά τη διάρκεια του 2008. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε επιτυχία αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του έτους και ήταν το ίδιο επιτυχή με τα προηγούμενα χρόνια και το προηγούμενο χρονικό διάστημα εν γέννη και είμαι βέβαιος ότι και η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι θετική. Επειδή τώρα μας πιέζει και λίγο χρόνος, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες και στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση και που ακούσαμε από τον κύριο Μέισταντ στην παρουσίασή του. Αυτό που σαφώς πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι η τράπεζα λειτουργήσε καλά και είχε πολύ καλά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του 2008. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια πράγματα, ότι πρέπει η Ευρώπη να έρθει πιο η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της, κυρίως σε περιόδους τις οποίες ε, είναι άμεσες οι επιπτώσεις ε, στους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί ε, μπορούν ίσως να διαπιστώσουν ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί μπορούν να έχουν κάποια επιρροή στην καθημερινότητά τους. Αν λοιπόν η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών είναι καθυστερημένοι, όπως για παράδειγμα των τραπεζών ε, για την έκδοση δανείων, ε, ή ορισμένες φορές είναι πιο γρήγορη η αντίδρασή τους όταν πρέπει να ζητήσουν καταβολή πληρωμών. Το 2008 λοιπόν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε ακριβώς το αντίθετο. Αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις χρηματοοικονομικής κρίσεως και όπως μπορούμε να δούμε και στην ετήσια έκθεση και ακούσαμε άλλωστε και στην παρουσίαση, η τράπεζα ενίσχυσε τις διαδικασίες δανεισμού και επίσης έλαβε και εξωτερική χρηματοδότηση για να μπορέσει να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, κατ' εξίσου σημαντικό, σαφώς δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ο τέλειος οργανισμός, το τέλειο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Άρα ούτε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι τέλεια. Όμως, Θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί πάρα πολύ σημαντικά βήματα για να ε, ενισχυθεί ο, ο ελεκτικός ε, ρόλος και να αυξηθεί η διαφάνεια, δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ετοίμασε κάποιες συστάσεις στο παρελθόν, οι οποίες κατά την άποψή μου είναι δικαιολογημένες ε, με βάση και τις δραστηριότητες της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Να γίνω λίγο πιο σαφής. Στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να βρούμε ποιες είναι αυτές οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν είναι δημόσιες σαφώς που μας αφορούν και προκύπτουν από τις δραστηριότητες της τράπεζας. Θα πρέπει να καθορίσουμε ποιε είναι αυτές οι δραστηριότητες, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα για να είναι πιο διάφανες οι διαδικασίες. Ε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι του δεν φαίνεται να οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις... ε, ε διαμαρτυρίες που είχαμε ως προς τη δραστηριότητα της τράπεζας. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτά τα στοιχεία και ε, να φροντίσουμε οι δραστηριότητες της τράπεζας να είναι όλο ένα και πιο διάφανες. Ολοκληρώνοντας λοιπόν να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για αυτή την έκθεση και ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα είναι ενημερωτική και ότι θα έχω και καλή συνεργασία με τους συναδέλφους ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Λούντμπορς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξάτομοι κύριοι βουλευτές. Σύντομα, θα αναφερθώ σε μερικά σημεία κάτι που το ανάφερε και ο ίδιος ο κύριος Μεστάντ. Η εποπτεία των τραπεζών. Όπως ξέρετε το συνέδριο δεν έχει εντολή γι' αυτό. Πάντως θεωρώ θετική τη δυνατότητα με την εποπτική αρχή της τράπεζας να έχουμε κοινέ δραστηριότητες να καλύψουμε δηλαδή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μια, να μπορεί να επεκταθεί η Επιτροπή από 3 σε 6 μέλη βάσει συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό είναι μια να είναι η, η, η απάντηση που ψάχνουμε. Κάτι άλλο που το ανάφερε επίσης ο κύριος Μεστάντ, η συζήτηση που θα γίνει για την εξωτερική εντολή της τράπεζας. Ευχαριστώ την προσοχή των ε, κυρίων βουλευτών. Όπως θα είδατε, το Συμβούλιο, το Συνέδριο έχει κάνει μια έκθεση σχετικά με τα μέτρα της τράπεζας ΜΕΔΑ 1, ΜΕΔΑ 2, και αυτό θα το συνεχίσουμε σαν σπάγια τακτική. Και παλιότερα σε εκθέσει δηλαδή το 2006 κοιτούσαμε κατά πόσον από νομική σκοπιά τηρήθηκαν όλοι οι τύποι για το ΜΕΔΑ 2. Έχουμε το κεφάλαιο 11 και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ανάφερε ο κύριος Μεστάτ για την συγκεκριμένη αντίστοιχη πολιτική της τράπεζας. Αύριο στην ημερήσια διάταξη έχετε την απαλλαγή για τα Ευρωπαϊκά Τιμή Ανάπτυξης. Το συνέδριο στην ετήσια έκθεση επεσήμενε ότι το εργαλείο επένδυσης κοτονού δεν τη αντικείμενο μελέτης εκ μέρους μας. Ενδέχεται όταν θα γίνει η αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών το 2010 να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ο Μπέρμα. Θα μιλήσω γαλλικά. σεβασμό προς τον πρόεδρο της τράπεζας, ο οποίος ο ίδιος μίγησε σε άριστα γαλλικά. Τον ευχαριστώ για την σαφή εισαγωγή του. Μία ερώτηση ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Εδώ είμαι να πληρωτήσω. και για το μέλλον της ε, Τράπεζα. Θα πάρει και μια έκθεση πρωτοβουλία. Γιατί προβλέπω λαμπρό ρόλο για την τράπεζα, για την ανάπτυξη στο μέλλον. Ερώτηση. Μιλήσατε για τους φορολογικούς παραδείσους. Μάλλον όρο βέβαια, αλλά αυτό εννοούσατε. Πρόσφατα εφαρμόζεται μια ενδιάμεση πολιτική σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έχουν βάση στους φορολογικούς παραδείσους. Έγιναν θετικά βήματα. Μιλήσετε όμως για ιδιώτες οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν τη βάση στους φορολογικούς παραδείσους. Τα χρήματα που δίνεται όμως σε τέτοιου είδους εργολάβους, από τη στιγμή που γίνεται το έργο, δεν, μπορείς, δεν μπορούν μετά να φύγουν προς φορολογικούς παραδείσους. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα χρήματα να μείνουν στη χώρα που έχει το πρόγραμμα. Διαφορετικά δεν ωφελούνται οι πολίτες Οφειλούνται κυρίως οι τραπεζίτες, οι χρηματιστές και οι ιδιοκτήτες και δεν είναι αυτός ο στόχος. Ένας από τους στόχους της Λισαβόνας είναι οι πολιτικές μας να μην παρουσιάζουν ανακολουθίες όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξη. Ερωτώ λοιπόν, τι μέτρα θα λάβετε έτσι ώστε τα χρήματα να μην φυγαδεύονται προς τους φορολογικούς παραδείσους. Είναι εξαπλάσιο το ποσό που φεύγει από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς τους φορολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, στο τέλος θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο μας Τάντη Χατζημαρκάκης. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα κύριε Πρόεδρε. Ακόμα και όταν τα λέω γερμανικά, σε πολύ ωραία γαλλικά μίλησε ο κύριος Μεστάτ. Εμείς είμαστε μόνο εμέρια αρμόδιοι. Ε, έχουμε και συναρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής αφενός και αφετέρου οι διοκτήτες της τράπεζας είναι τα κράτη-μέλη. Και βέβαια με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε ενισχυμένο ρόλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να επενέσω πάρα πολύ το, το ρόλο της τράπεζας στην χρηματοοικονομική κρίση. Πάντα είχατε φρόνιμη και συνετή διαχείριση και μπορέσατε να βοηθήσετε γιατί δεν σας έπληξε η κρίση. Καλούμε να το διαπιστώσουμε αυτό και, και ε, Ευρωπαίοι ε, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τη δική μας τράπεζα, γιατί είστε η δική μας τράπεζα, η μεγαλύτερη τράπεζα επενδύσεων στον κόσμο. Τώρα εγκρίναμε ένα σχέδιο ανάκαμψη και πολύ γρήγορα πρέπει να τεθούν σε ισχύ τα έργα. Εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί με δύο-τρία έργα και μίλησα και με μέλη τη Τράπεζά σα και η συμπεριφορά του δεν ήταν μόνο ορθή και ε, άψογη, αλλά ήταν και ταχύτατη ανταπόκριση και πρέπει να το πούμε αυτό. Σε αυτό το πρόγραμμα για την ανάκαμψη μπορούμε να βασιστούμε πάνω σας και τα πολιτικά θέματα που έχουμε βάλει στην ημερήσια διάταξη, ιδιαίτερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα τα εφαρμόσουμε κιόλας με τη βοήθειά σας. Από το παρελθόν μπορώ να σας πω, όχι μόνο για την τράπεζα, γιατί είστε και όμιλος, έτσι, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, κάθε φορά που χρειάστηκε να συνεργαστώ μαζί τους, ω εισηγητή, για το πρόγραμμα πλαίσιο για την κοινοτομία δεν έχω παρά επένους να πω και καλά λόγια. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ομαλά, με πολύ μεγάλη διαφάνεια όπω και η έκθεση δραστηριοτήτων και πεπραγμένων σα ε, για την εταιρική ευθύνη, κοινωνική ευθύνη, το διαπιστώνουμε. Είστε ένα όργανο πάρα πολύ ανοιχτό, με διαφάνεια και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Έχω τώρα μια-δυο ερωτήσεις ε, για το μελλοντικό σα ρόλο για τις εξωτερικές δραστηριότητε. Από το 2010 και μετά, το είπατε κι εσείς ο ίδιος και το εξηγήσατε, έχετε νέο πεδίο εντολής και ορισμού των εντολών και θέλω να ρωτήσω εκεί πώς σκοπεύετε να αποφύγετε την επικάλυψη. Υπάρχει στο Λονδίνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Ξέρω ότι επιτέλους θα έχουμε ένα γενικό σχεδιασμό του τραπεζικού τοπίου, του ευρωπαϊκού εννοώ, και πώς ε, θέλετε να ε, αποφύγετε αυτές τις επικαλύψεις με την BERT. Μετά, έχουμε τη Βαρόνη Άρστον πλέον. Είπα ότι εκπρόσωπο πώς αλλάζει η ύπαρξή της και μόνο και η ανάληψη καθηκόντων της το δικό σας ρόλο. Γιατί και εκεί υπάρχει νέα όθηση. Μιλώ πάντα για τις εξωτερικές δράσεις. Πώς θα επηρεαστούν αυτές και πώς θα αλλάξουν και πολύ συγκεκριμένα τι εστί ευρωπαϊκό συμφέρον. Ακούω ότι δραστηριοποιείται σε μεγάλα έργα η τράπεζα παγκοσμίω όπου δεν έχουμε καθόλου ευρωπαϊκή συμμετοχή. Εντάξει, η δική σας εποχή στο γιατί υπάρχουν και ανταγωνισμοί παγκοσμίω. Είναι ε, προϊόντα με πρώτε ύλε, όπου τελικά κάπου στο τέλος οι Ευρωπαίοι εποφελούμαστε. Αλλά άμεσο συμφέρον δεν βλέπω και άμεσο όφελο και άμεση σχέση. Και είναι και γενναία χρηματοδότηση εκεί. Εσείς είστε πρόθυμοι να βρούμε ένα κοινό ορισμό του ευρωπαϊκού συμφέροντος και προς το σκοπό αυτό να κάνετε τα δανειά σας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη συνάδελφε. Φτάσαμε στις 6.30. Πρέπει να κλείνουμε και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μεσταντέ. Έχουμε τέσσερις συναδέλφους. Σας παρακαλώ ένα λεπτό ο καθένας να σας δώσει το λόγο γιατί ο πρόεδρος έχει έρθει και θα ήθελα να μιλήσει τελευταίος. Μπάλτσιντης. Ačiū labai gerimas pirmininkė dėl Europos investicinio banko. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά ωραία λόγια για την τράπεζα και είχα την ευκαιρία να με την τράπεζα στη χώρα μου όταν ήμουνα υπουργό Οικονομικών. Η κατάσταση όμως άλλαξε. Μη θλίψη μου, μάλλον είναι ατυχές, αλλά πρέπει να μιλάμε για ορισμένες χώρες μέλη που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Αναφέρεται τις χώρες της Βαλτικής. Έχουν προγράμματα ενεργειακά για την ε, αναπαλαίωση κτηρίων, εξυγχρονισμό κτηρίων. Και ακούμε ότι ορισμένα προγράμματα προς χρηματοδότηση παρά είναι γραφειοκρατικά. Πριν έρθει κύριε Πρόεδρε, συζητούσαμε εδώ ότι πρέπει να μειώσουμε την πολυπλοκότητα των κανονισμών. Το επισημαίνω αυτό. Πρόεδρος ο ο Ντί. Μερικά μικρά σχόλια. Μπορείτε να μας πείτε κύριε Πρόεδρε δύο λόγια για την ε, ποικιλομορφία των αποτελεσμάτων σας το 06 3 δις μετά κατεβαίνουμε στα 8, ε, συγνώμη, 1 δις, 800 εκατομμύρια μετά έχουμε ε, σε 9 λογαριασμού 6 λόγω της αλλαγής των ισοτιμιών. Μεγάλες διακοιμάνσεις. Για να καταλάβω πού φύλλονται αυτές οι διακοιμάνσεις, οι αιτήσει. Για τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε την νομική, το νομικό πρόσωπο πια της Ένωσης. Η Ένωση θα μπορούσε να γίνει μέτοχος της τράπεζας επιπλέον των κρατών μελών. Χαίρομαι που είπατε ότι είστε ευρωπαϊκό εργαλείο και όχι διακυβερνητικό. Και τελευταίο, στην έκθεσή μου του 2006 ζήτησα η Κομισιόν να σας αναθέσει ένα είδος engineering για τη χρηματοδότηση. Δεν νομίζω ότι σας δόθηκε αυτή η εντολή από την Κομισιόν. Μας λείπουν εργαλεία επενδύσεων. Γιατί εσείς ως τράπεζα θέλετε να κρατήσετε το 3α που έχετε. Θα ήταν χρήσιμο αυτή η μελέτη. Γιατί νομίζω δεν επενδύει αρκετά η Ένωση. Πρόεδρος Αγιάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για τις ε, πληροφορίες και να ρωτήσω κάτι για το Ταμείο Μαρκερίτο που νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως ε, ασχολείται με τα θέματα αυτά. Είναι για μια πολύ... Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό όμιλο που ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Θα μπορούσατε να μα πείτε κάποια παραπάνω πράγματα. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο, διότι ξέρω ότι θέλετε να τελειώνουμε. Νωρίτερα κάναμε κάποια συζήτηση για την πολιτική συνοχή σε σχέση και με την έκθεση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου που συζητήσαμε νωρίτερα. Ξέρουμε όλοι ότι η πολιτική συνοχή είναι υπό απειλή και υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν ε, σε νέους ε, μηχανισμούς για το μέλλον, ε, ο μηχανισμοί όπως ο Τζέρεμι, ο Τζέρεμι και η Τζέσικα. Θα ήθελα οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να σχολιάσουν ε, τι θα γίνει με αυτά τα μέσα και τι μηχανισμούς θα έχουμε για να τα ελέγχουμε αυτά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο Μάισταν. Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις. Αν θέλει να μας πει κάποια πράγματα πιο διεξοδικά θα μπορούσε ίσως να μας τα αποστείλει γραπτός αν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντω, ακολουθήσω τη συμβολή σα γιατί είναι τόσε ενδιαφέρουσε ερωτήσει που θα άξιζαν βαθύτερη απάντηση. Τηλεγραφικά τώρα θα αναφερθώ επιγραμματικά και θα ακολουθήσουν ε, εκτενέστερε γραπτέ απαντήσει. Τώρα, για τα αποτελέσματα. Ο εισηγητής σας, ο κύριος Ντότς, ε, είπε και σημείωσε ότι πολύ λίγο μας επηρέασε η κρίση, γιατί με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο είχαμε κάνει τις επενδύσεις μας, παρά τις αιτήσει που δεχτήκαμε να ε, επενδύσουμε σε συγκεκριμένα προϊόντα που μας ζητούσαν επειδή το έκαναν όλοι οι άλλοι. Ανηθήκαμε και ευτυχώς αυτό ε, μας επέτρεψε να έχουμε αποτελέσματα και δεν μας επηρέασε τόσο πολύ η κρίση. Υπάρχει το πρότυπο EFRS, το διεθνέ. και τα πρότυπα αυτά ε, ενθαρρύνουν την πτυτικότητα και έπαιξαν ένα ρόλο προκυκλικό για την χρηματοοικονομική κρίση. Αν δείτε όμως ε, τους κανονισμούς και το καταστατικό μας και, τα, και ε, τους λογαριασμούς μας, τους ευρωπαϊκούς, ήταν 1 δις το 2008 και φέτος 1,7 δις ε, κέρδη. Δηλαδή αυξάνουμε σταθερά, αργά αλλά σταθερά τα ετήσια κέρδη μας. Δεν θα σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριος Λίμπορτς, αλλά γνωρίζετε ότι οι περισσότερες δράσεις μας είναι από πόρους που συλλέγουμε στις παγκόσμιες χρηματαγορές για το μικρό τμήμα που χρησιμοποιούμε δύο σπόρους ή από το κοινοτικό προπολογισμό είναι φυσιολογικότατο να μας ελέγχει το ελεκτικό συνέδριο. Και το κάνει. Βάσει ε, της τριμερού συμφωνίας που έχουμε για διάφορα σημεία έχει κάνει πολύ εύστοχες παρατηρήσεις στο ελεκτικό συνέδριο που πολλές φορές επιβεβαίωναν ε, τις βάσιμες αντιδράσεις ορισμένων, όπως ε, είπαμε τις ε, δράσεις για τη Μεσόγειο. Είπε το ελεγκτικό συνέδριο μερικά πράγματα και εμείς καταγγείλαμε και την παρακολούθηση του ελέγχου ήδη. Δηλαδή ήδη από το 2005 το είχαμε συνειδητοποιήσει και είχαμε λάβει μέτρα για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ο κύριος Μπέρμαν έκανε μια σημαντική όσο και λεπτή ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο εμποδίζουμε ε, τα κέρδη από μια χώρα να μην φύγουν προς φορολογικούς παραδείσους. Και αυτό μας απασχολεί, αλλά δεν είμαι πεπισμένος ότι η πολιτική που υιοθετούμε και είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον G20 και τις συστάσεις τους, είναι τελείως αποτελεσματική από αυτή τη σκοπιά. Και μας προβληματίζει αυτό και εξακολουθούμε να το μελετούμε. Ο κύριος Χατζημαρκάκης έκανε μια βασική ερώτηση και θεμελιώδη και θα πρέπει να επανέλθουμε στη συζήτηση αυτή για τις νέες εντολές για τις εξωτερικές δράσεις. Πώς ορίζεται το ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον. Απαντώ ξεκάθαρα στον κύριο Χατζημαργάκη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι απολύτως πρόθυμη να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη προβολή και ορατότητα και αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής δράσης. Γιατί σε πολλούς τομείς μόνο μέσα από το συνδυασμό ε, δανείων δικών μας και χρηματοδότηση από τον προπολογισμό έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και απόδοση μεγαλύτερη. Και αποτελεσματικότητα δηλαδή. Ήδη υπάρχει μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να διευρυνθεί και επανέρχομαι στην ερώτηση του κυρίου Οντή. Ένα τρόπο να ενισχυθεί αυτή η δυστενή και απαραίτητη συνεργασία ε, τη Κομισιόν με την τράπεζά μα είναι να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι άμεσα μέτοχο είτε τη ΕΤΕΠ είτε μια θηγατρική τη που ε, δραστηριοποιείται περισσότερο στο εξωτερικό. Θα επανέλθουμε σίγουρα όμω σε αυτά τα θέματα για την επένδυση που τράβηξε την προσοχή και του κυρίου και της κυρίας Αγιάλα Σέντερ μπορώ να σας πω για τη Μαργαρίτα αύριο τελειώνουμε την πρώτη φάση αυτού του ταμείου που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πανευρωπαϊκό ταμείο και έχει στόχο να φέρει κεφάλαιο ή σχεδόν κεφάλαιο σε μεγάλα έργα υποδομής τη ενέργεια και στι μεταφορές. Έξι ίδρυτες είναι η ίδια η τράπεζά μα, η ΣΕΝΤΕΣ γαλλική, η ε, ε, ιταλική, μία υπό, από την Ισπανία, ΠΕΚΑ, Πολωνία και μία γερμανική τράπεζα. Αλλά βεβαίως παραμένουμε ανοιχτοί σε άλλες συμμετοχές, σε άλλους επενδυτέ, Αύριο θα ξεκινήσουμε εμεί. οι έξι καθένα βάζει 100 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με κάποιου άλλους μέχρι τα τέλη του έτου θα φτάσουμε στα 750 και έτσι θα αρχίσουμε την προσπάθεια αυτή και υπάρχουν κάποια έργα που δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται αμυγός από ε, δάνεια για να έχουμε και μετοχικό κεφάλαιο. Και προς τον κύριο Βόγκα να απαντώ στα αγγλικά. Ε, θα σας ενημερώσω πάρα πολύ σύντομα θα σας στείλω περισσότερες λεπτομέρειες γραπτός για την Τζέσικα και τον Τζέρεμι. Τα νέα μέσα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον Τζέρεμι η ιδέα είναι να μετατραπούν τα διαρθρωτικά ταμεία κονδυλία σε δύο ανανεώσιμα μέσα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων και θα σας δώσω τον αριθμό συμφωνιών που ήδη έχουμε συνάψει ε, στο Τζέρεμι και η Τζέσικα είναι η ίδια ιδέα. Ε, μετατροπή των διαρθρωτικών πόρων σε συμμετοχή σε ταμεία αστική ανάπτυξη, δηλαδή αστική ανοικοδόμηση, ανανέωση των πόλων, αναζωγόνησης. Είναι πιο πρόσφατο, μόλι τώρα ξεκινάει, αλλά έχουμε ήδη ολοκληρώσει κάποιε συμφωνίε και προγραμματίζουμε και άλλε. Θα σα ενημερώσω σε λεπτομέρειε γραπτός για το πού βρισκόμαστε με τα δύο αυτά έργα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Επειδή είναι πολύ χρήσιμη η συνεισφορά σας, έλεγα λοιπόν ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Περιμένουμε και κάποια γραπτά στοιχεία για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτά που μόλις μας είπατε. Ναι, μεν τα εξαντλήσετε τα θέματα, αλλά επειδή τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερως ευαίσθητα, ε, ίσως πρέπει να λάβουμε και τα γραπτά σας. Καλό λοιπόν στη μικρή δεξίωση. Είστε